Colleagues, if I could reconvene the meeting, Ξεκινούμε, συνάδελφοι. Σας παρακαλώ. Ξεκινώ με τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου μετά την συνάντηση των συντονιστών χτες. Πρώτον, εγκρίθηκε το σχέδιο υπηρεσία διάταξης και μετά εξετάσαμε την εντολή διαπραγματεύσεων για τα τέντη παρουσία των εισηγητών κ. Κουμουτσάκου και ε, Τούγκ. Η απόφαση των συντονιστών ήταν να συστήσει στην Επιτροπή να αποφασίσει, ήταν απόφαση με πλειοψηφία, για να ξεκινήσουν οι άτυπες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με βάση την ε, εντολή της έκθεσης που υιοθετήθηκε στην Επιτροπή και με την ε, διαπραγματευτική ομάδα που θα περιλαμβάνει τον πρόεδρο, τους εισηγητές και τους κοιόδης εισηγητές. Η απόφαση θα ληφθεί, η επίσημη απόφαση θα ληφθεί σήμερα. Για το πακέτο αεροπορικών μεταφορών παρουσία του εισηγητή κ. Ζασάντα αποφασίστηκε να οργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ εισηγητού και σκιωδών εισηγητών τη Επιτροπή Μεταφορών και τη Επιτροπή Απασχόληση στο Συνωμό των Δεντών για να προσπαθήσουν να λύσουν τι δυσκολίε που υφίστανται. Για το πακέτο των σλότ τώρα αποφασίσαμε να μείνει ω πακέτο στη φάση αυτή μαζί με, το με την πρόταση για το ground handling παρότι αναγνωρίστηκε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία για το ground handling θα πρέπει να επανέλθουμε. ισμός εισηγητών πρόταση κανονισμού για τις, ε, την, τις αναφορές στην πολιτική αεροπορία. Η ΕΛΚ θα δώσει εισηγητή. Πρόταση οδηγίας για τον ε, εξοπλισμό, ένα άλλο εξοπλισμό που καταργεί τον, κανονισμό 96-98. Δεν το ήθελε καμία ομάδα το κείμενο αυτό, αλλά ο πρόεδρος δεν αναλάβει την έκθεση. Γνωμοδοτήσεις. Η πρόταση του, του κανονισμού Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό 994 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης σε, ορισμένο ε, σε ορισμένο των ε, κρατικών ενισχύσεων κανονισμού 1370 των υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών οδικά και συνοδομικά. Θέμα κρατικών ενισχύσεων στις δημόσιες μεταφορές, τομέας των οποίων υπήρχαν κάποιες ανησυχίες της Οικονομικής Επιτροπής, της κύριας Επιτροπής. Η απόφαση των συντονιστών είναι να σας προτείνει να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 50. Ο πρόεδρος να λειτουργήσει ως εισηγητής είναι ένας τομέας αλλά σημαντικός για μας. Ανα... Άλλη γνωμοδότηση για την ανακοίνωση ενίσχυσης της ενίας αγοράς ε, καταργώντα, ε, αφαιρώντας τις, ε, φορο, τις επιφορολογικές των επιβατικών αυτοκινήτων. Η ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η ανακοίνωση για την έκθεση ποιότητας των, ε, του ντίζελ οδικών μεταφορών και για τους τελικούς, τον τελικό απολογισμό της Ένωσης 2011 αποφασίστηκε να μην γίνει δράση ούτε και να υπάρξει δράση για την κοινή ανακοίνωση υπέρ της στενότερης συνεργασίας μεταξύ ε, και την περιφερειακή ενοποίηση στην περιοχή του Μαγκρέμπ. Ούτε εδώ υπάρξει ε, πρόταση. Οι συντονιστές εξέτασαν το θέμα της ασφάλειας των εναέριων μεταφορών ιδιαίτερα την έκθεση ε, της, το ρόλο της ΙΑΣΑ μετά το ατύχημα του Κονκόρντ καθώς και τις ασφ, συνθήκες ασφάλειας για τα επίπεδα καυσίμων και τα λοιπά στις εταιρείες χαμηλού κόστους. προτείναμε να ζητήσουμε από την ΕΑΣΑ να έρθει σε μια μελλοντική μας συνάντηση για να το συζητήσουμε. Επίσης εξετάσαμε κατά πόσον υπάρχουν επιπτώσεις ασφάλειας ε, λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης για τις αεροπορικές μεταφορές στην Ένωση. Επόμενο θέμα. Η πρωτοβουλία της ΙΜΚΟ για μια νέα ε, ημερήσια διάταξη για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών. Αποφασίστηκε ο πρόεδρος να στείλει επιστολή στην, στον πρόεδρο της ΙΜΚΟ. Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του 2013 σας το στείλαμε. Άλλαξε, όπως ξέρετε, η ημερήση, άλλαξε το πρόγραμμα μας λόγω της δεύτερης συνάντησης ε, ολομέλεια τον Οκτώβριο που συμπίπτει με συνάντησή μας. Αναθεωρήσαμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα, δείτε το, δείτε τι σας ζητούν, ε, με τι σα ζητούν να συμφωνήσετε οι συντονιστέ. Επί τροπολογία σημειώσαν ε, οι συντονιστέ ότι οι εσωτερικέ προθεσμίες της ΙΚΟ έληξαν χωρίς, χωρίς η προθεσμία είναι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσημες προτάσεις για τον περιορισμό των ε, πτήσεων. Η άποψη των συντονιστών είναι να έχουμε ακρόαση για το θέμα αυτό. Σας το λέω διότι είχαμε σήμερα διαδηλώσεις, όπως και το Κοινοβούλιο ωστόσο δεν έχει θέση γιατί δεν λάβαμε επίσημη θέση από την Επιτροπή. Κάθε απόφαση σχετικά με τον χρόνο, με τη διάρκεια πτήσεων και τη διάρκεια ε, υποχρώσεων των ε, ε υπαλλήλων ε, στηρίζεται στο ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να πει ναι όχι, δεν μπορεί να σχολιάσει κάτι. Διάφορα, ε, τα διάφορα. Το, ατύχημα Φλαμίνια. Θα απαντήσει ο πρόεδρος στην Επιτροπή του κ. Κάλλας ε, που ζητούσαμε περισσότερες πληροφορίες από την αρχική απάντηση. Για τα τεράστια πλοία τώρα, τα gigaliners, δεν τα τεράστια οχήματα, τα gigaliners συγγνώμη, η απόφαση την περασμένη εβδομάδα ήταν ε, να ζητήσουμε από τον πρόεδρο Σούλτς να στείλει επιστολή στον πρόεδρο Μπαρόζο για να προσπαθήσουμε πώς το πω τώρα να μειώσουμε την σύγχυση που προκύπτει από την απάντηση της Επιτροπής στην γενική συζήτηση. Αυτά από τους συντονιστές. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. Κύριε Λιμπεράτσικη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εξετάσατε το τεστ, το, είδατε καθόλου συντονιστές το τέταρτο πακέτο συνδεδομικών μεταφορών. Διάβασα το κείμενο και έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος της Deutsche Bank, της Deutsche Bahn θα ζητούσε από την κυρία Μέρκελ να αποφασίσει ε, που σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε πια πακέτο. Έχουμε μεγάλες ε, καθυστερήσεις στην παροχή των κειμένων από την Επιτροπή. Μας είχαν υποσχεθεί στις 17 Δεκεμβρίου πρώτα μας στείλουν τα κείμενα, μετά μας είπαν 15 Ιανουαρίου. Μήπως θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να επιταχύνει την υποβολή του πακέτου γιατί αλλάζουν πράγματα. Δεν συζητήθηκε το θέμα αυτό στον, στους συντονιστές. Ξέρω ότι η Επιτροπή ζήτησε να περιμένουμε μία εβδομάδα τους ώστε ο πρόεδρος ε, να πάει στο Βερολίνο να μιλήσει με την κυβέρνηση της Γερμανίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε στη φάση αυτή. Η Επιτροπή ε, περιμένουμε για την Επιτροπή. Αν, το, υπάρξει πρόβλημα και μετά την επιστροφή από, την, ε, από το Βερολίνο, θα μας κάνει πρόταση η Επιτροπή και θα αναλάβουμε και εμείς δράση. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή το σωστότερο θα ήταν, παρά την καθυστέρηση, το σωστότερο επαναλαμβάνω θα ήταν να δώσουμε στην Επιτροπή μια εβδομάδα ακόμα για να μιλήσει με τη γερμανική κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Εντάξει. Δεκτή, έτσι. Προχωρούμε. Ψηφοφορίες. Κάντε ένα, κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε αν όλοι είστε έτοιμοι. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για να κάνουμε έλεγχο. Κάποιος άλλος ξέρει σε κάρτα. Ωραία. Αν με το καινούριο χρόνο να πω ότι δεν είστε περισσότεροι από το ΕΛΚ σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Καλά ξεκινάμε. Αυτό ως χωριστό πρακτικό. Ξεκινούμε. Γενικός προϋπολογισμός, απαλλαγή 2011, τμήμα 3. Επιτροπή. Η κυρία Ντιρόν, η Υπάρχει μια προφορική τροπολογία της εισηγήτριας που αντικαθιστά την παράγραφο 1, την έχετε. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία, αν όχι, θα μπούμε με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή Δύο. υπέρ κατά αποχές δεκτή Τρία. υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας 36 υπέρ, 2 κατά 2 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Επόμενη έκθεση. Σχέδιο γνωμοδότησης για την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ΕΜΣΑ. Προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών υπάρχει. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Αν όχι, θα τη συμπεριλάβουμε. Τροπολογία 1 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για το τελικό κείμενο. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 38 υπέρ, 2 κατά, συγχαρητήρια. Κυρία Μάισνερ, εγκρίνεται. Εάσα. Απαλλαγή πάλι. τις κυρίες Μέισνερ. Της τροπολογία 1. Τάντι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2. Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Όχι. Με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. 37 υπέρ 3 κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι. Ζεζίν. Επόμενο. Της Ζεζίν πάλι. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία με τροπολογία 3 υπάρχουν αντιρρήσεις αν όχι 3 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 37 υπέρ 3 κατά. Συγχαρητήρια και πάλι προς την κυρία Μάισνερ. Γκρίνεται. Σεζάρ. Κοινή επιχείρηση Σεζάρ. Απαραγή 2011. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τρία τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Ζεζίν για όλες τις εκθέσεις. Επόμενο. Έκθεση δύο πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού. Ο κ. Καμάλιν είναι εισηγητής. Τροπολογία 1. Υπέρ. Μαζί τροπολογία 1 και 2, έτσι. Μισό λεπτό. Όχι. Ψηφίζουμε χωριστά και μετά θα συνενωθούν αν γίνουν δεκτές. Τροπολογία 1. Κράμερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 με κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπογραμμίζει για τις μεταφορές υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα καλή κλπ υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές έλεγχος έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την τοπολογία 10 ψηφίσετε όλοι πέρα ψηφοφορία. απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17. Τίκαο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Το τελικό τμήμα της 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21. With a view to making. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 28 άρχητη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τριάντα δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Να μου λένε ότι το ΕΛΚ είναι ένας παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30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 Πέρας ψηφοφορίας. Ε, δεν νομίζω χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Ρικέ. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 39. Μπένιον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απολύπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 είναι προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 καταπίπτει, 44 καταπίπτει και 43 καταπίπτει. Στη 44 υπάρχει μια προσθήκη. Τι... No, no, they all, they, they fall, they fall because it's not. Καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε 42. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα 40 αποσύρθηκε λόγω της προφορικής σαράντα 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Γιατί 46 ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 47 πρώτο τμήμα μέχρι το πατήσιμο της Ιζενσού. Υπέρ. Κατά. Ξανά. Για το 47. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα γίνει ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για το 47. Ψηφίσετε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 48. Διοθώνει ο πρόεδρος. Το δεύτερο τμήμα του 47. Το δεύτερο τμήμα του 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το 12 καταπίπτει φαντάζομαι παρότι είναι μόνο το ένα. Τμήμα 48 υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας 36 υπέρ 3 κατά εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Καμάλ. Επόμενο θέμα. Ξεκίνημα διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής για το δίκτυο TNT. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρα ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 6 άρα εγκρίνεται η εντολή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν κυρίες και κύριοι και έτσι ελευθερώνουμε τις ψηφοφορίες μας. We now go on to Aviation ETS Stop the Clock, consideration of the draft opinion of Mr. Grosh. Matthew on floor. Κοιτάξουμε λοιπόν τώρα την εκτέλεση του κυρίου Grosh. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Στο θέμα αυτό έχουμε λίγο ε, χρονική πίεση. Παρόλα όλα αυτά όμως θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε σωστά αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε πλέον μιλάμε για τις πτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, να επεκταθεί δηλαδή και σε αυτές τις πτήσεις, αν και ξεκινήσαμε από το 98 να αναζητούμε λύσεις για το παγκόσμιο αυτό πρόβλημα, παρουσιάζονται προβλήματα ακόμα, αλλά στην συνάντηση το Νοέμβριο σημειώνονται θετικά στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν και γίνεται αυτή η πρόταση. Καλωσορίζω λοιπόν την προσέγγιση αυτή και νομίζω το έχουμε πει και στο παρελθόν. Αυτή η αρχή του ETS ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Απλά θέλουμε να δώσουμε την ε, ευκαιρία να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζει αυτή την επέκταση προσωρινά σε ένα έτος. Σε διάφορες τροπολογίες σημειώσαμε με σαφήνεια ότι για μας πρόκειται για ένα έτος. Και θέλουμε φυσικά να δούμε και τι θα γίνει, ποια θα είναι τα αποτελέσματα ε, του 2013 και ότι θεωρούμε ότι αν δεν έχουν σημειωθεί πρόοδοι μέχρι τότε, θα επανέλθουμε στην ισχύουσα νομοθεσία και το ETS ε, θα, χρησιμο... θα εφαρμόζεται χωρίς περιορισμό σε όλες τις πτήσεις. Αλλά εάν η ΚΑΟ αν ε, διαφανούν κάποιες επιτυχίες ε, του συστήματος αυτού, θα θέλαμε να ενημερώσει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Κοινοβούλιο με πλήρη διαφάνεια, καταρχάς, και κατά δεύτερον, προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβεί σε περαιτέρω βήματα και φαντάζομαι ότι αν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, θετικά πορίσματα, ε, θα είναι απαραίτητο να κάνει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε δύο σημεία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Καταρχάς, ε, να μην λαμβάνονται μέτρα τα οποία θα στρεβλώνουν την αγορά, δηλαδή να ισχύουν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να ισχύουν σε διεθνές επίπεδο κτλ. Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και κατά δεύτερον η συζήτηση θα πρέπει να ε, ε, ενέχει και στην συζήτηση θα πρέπει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στο μέλλον. Κοιτάξτε, είναι λίγο ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μα, αλλά δεν είναι και αδύνατον να τα ολοκληρώσουμε. Η ΕΝΒΗ παραμένει η καθήλυνα αρμόδια. Συνεχίζει συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε, γνωμοδοτούμε απλά. Θέλει η ΕΝΒΗ στις 26 να ψηφίσει την έκθεση αυτή, άρα και εμείς να θέσουμε ανάλογες ε, καταληκτικές ημερομηνίες για τις τροπολογίες για να μπορέσουμε να δώσουμε την οικονομοδότηση και να τη λάβει υπόψη η ΕΝΒΗ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκρός, ο κύριος Ελκαντράουι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισήγητη για τη γρήγορη δουλειά που έκανε πρέπει να τοποθετηθούμε ως επιτροπή και διαπιστώνω ότι σήμερα δεν απέχουμε τόσο πολύ από την κατάσταση την οποία είχαμε προτείνει εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών όταν καταρτίστηκε πριν από δύο χρόνια η νομοθεσία που είχαμε πει να δουλέψουμε σε δύο βήματα. Δηλαδή στην αρχή να ε, εφαρμοστεί το σύστημα εκπομπών ρήπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε μετέπειτα φάση όταν θα έχει δουλέψει λίγο το σύστημα και όταν θα έχουμε συζητήσει το σύστημα αυτό με τις άλλες ε, χώρες να το επεκτείνουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Ο νομοθέτης ε, τότε αποφάσισε διαφορετικά και ξέρουμε τι δυσκολίες ε, προκλήθηκαν. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι είναι καλή και λογική. Ας αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτό το άνοιγμα που μας δίνεται σε ό,τι αφορά και την συνάντηση της ΙΚΑΟ όπου εκφράστηκε μία δέσμευση για μια, ένα σχέδιο πρότασης για μια παγκόσμια λύση. Κοιτάξτε, ή θα πετύχει αυτό και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Είτε θα αποτύχει και θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιμείνουμε η νομοθεσία η οποία έχει εγκριθεί ασφαλώς και θα πρέπει να γίνει σέβαστη και μια άλλη ενδεχόμενη λύση είναι να σημειωθεί μια πρόοδος αλλά να μην υπάρχει μια τελική συμφωνία, να πρέπει να διευκρινιστούν ακόμα λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν ε, πρέπει τώρα να το αναφέρουμε αυτό ως ενδεχόμενη λύση, γιατί ίσως να αποδυναμώσει την θέση μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να το σκεφτούμε, δεν ξέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απολύτως απαραίτητο στο ενδιάμεσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους μήνες ε, να ενημερώνει την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο για τις σχετικές εξελίξεις προκειμένου να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε οριστικά. Thank you, Mrs. Meissner. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να πω μετά από αυτά που είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητέ. Όντω, έκανε μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έχει τοποθετηθεί. Είμαι αισιόδοξη. Ελπίζω να υπάρξει μια παγκόσμια συμφωνία Ασφαλώς δεν θα είναι το ίδιο το πρόγραμμα ETS, πρόγραμμα ανταλλαγής ρήπων. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αλλά αν δεν προκύψει συμφωνία, Κοιτάξτε, πάντα ήταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει το παράδειγμα στον τομέα αυτό. Τόσο που σκεφτήκαμε και μήπως προκαλείται στρέβλωση για τις δικές μας αεροπορικές εταιρείες. Γι' αυτό λοιπόν η κατάσταση είναι δύσκολη. Επαναλαμβάνω, μακάρι να καταφέρουμε να περάσει σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή η συμφωνία, γιατί αυτό θα ήταν φανταστικό, θα εξυπηρετούσε και με το βέλτιστο τρόπο τον σκοπό μας, το στόχο μας. Να παρακολουθούμε λοιπόν στενά την κατάσταση και θα πρέπει όντω η Επιτροπή να μας ενημερώνει. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ. Ναι, υποστηρίζουμε την έκθεση επί της αρχής, την έκθεση του κυρίου Γκρός. Τι είναι όμως σαφές ότι το trading system, το σύστημα εμπορίας ε, δικαιωμάτων εκπομπής δεν εκπληρώνει τους στόχους ε, που είχαμε θέσει στην... Ε, μιλάμε τώρα για 5 ευρώ. Στην αρχή μιλούσαμε για 10-13 ευρώ. Θέλαμε να υπάρχει ανταγωνισμός. Πλέον όμως δεν υπάρχει ανταγωνισμός, έχει καταργηθεί ουσιαστικά. Είναι η τελευταία ευκαιρία να εφαρμοστεί αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά είμαι μάλλον απεσιόδοξο, γιατί οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, λένε ότι ναι, να συμφωνήσουμε αρκεί να υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις στην Ευρώπη. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο Β όταν εισήχθη το σχέδιο εμπορίας ρήπων, το αποτέχθηκαν οι αεροπορικές γραμμές επειδή φοβούταν ότι θα υπήρχε ε, φόρος επί της κυροζήνης. Φυσικά, αν υπάρξει τέτοιο φόρος, θα κρυβίνουν οι πτήσεις συνολικά και αυτό θα είναι ένα περαιτέρω βήμα για την εσωτερικοποίηση των εξωτερικών, του κόστους. Αλλά πάντα υπάρχουν ε, δισταγμοί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Αυτό θα ήταν το επόμενο βήμα και η απαλλαγή από το φόρο κυροζήνης δεν είναι κάτι που ισχύει παγκόσμιο. Κάποιες ε, χώρες επιβάλλουν τέτοιο φόρο. Αυτό θα ήταν για μένα το σχέδιο Β. Γιατί οι αερομεταφορές είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, δεν μπορούν να συνεχίσουν ε, όπως είναι σήμερα. Θα μπορούσαμε να δείξουμε λοιπόν και στους άλλους, γιατί είναι ισχυρό παράγοντας η Ευρώπη με 550 εκατομμύρια ε, καταναλωτές, ότι έχουμε δύναμη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τα έχουμε αυτά στο πίσω μέρος του μυαλό μας και να το ξέρουν και οι άλλοι. Δεν θα τη γλιτώσουν δηλαδή χωρίς έξοδα. Μπορεί, άμα δεν συμφωνήσουμε, τελικά να χρειαστεί να πληρώνουν και περισσότερα. Γιατί ξέρετε ότι οι εκπομπές είναι εξίσου επικίνδυνες και στη στρατόσφαιρα όσο και στη δική μας την ατμόσφαιρα. Φανώς ε, δημιουργούμε στις αερομεταφορές ε, μία φούσκα, όπως τα ακίνητα. Και αυτό οδηγεί σε ε, μεταρρυθμίσεις, σε αλλαγές στα αεροδρόμια και αυτά τα πληρώνει ο φορολογούμενος και δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να την πληρώνει ο φορολογούμενος, γιατί θα πρέπει να χρηματοδοτεί ο φορολογούμενος. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. thank you, Chairman, and um, uh, huge thanks to... Uh, ήθελα να ευχαριστήσω τον Ματιού για την έκθεσή του. Νομίζω ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέσο και προφανώς φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να ιτιές το σύστημα αυτό να το καθυστερήσουν και πιστεύω, νομίζω ότι θα πρέπει η θεσμή αυτή να ισχύσει για όλες τις τήσεις. Δεν θέλουμε να επικρίνουμε για αυτό το θέμα την Γενική Διεύθυνση μου, διότι Λάχισαν από την ΕΜΒΗ και τώρα προσπαθούν οι πάντες να δουν τον μπέρδεμα που είχε δημιουργηθεί πώς θα μπορέσει να το ε, επιλύσουμε. Δεδομένου ότι δεν είχε εκπλήσει κανείς περίπτωση πρόκειτο καταρχάς. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε τα κατάλληλα μέτρα για όλες τις μορφές μεταφορών και για όλη τη σχετική βιομηχανία που είναι υπεύθυνη για την εκπομπή αερίου. αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά ε, δημιουργήθηκε μια μεγάλη σύγχυση παγκοσμίω και σε πολιτικό επίπεδο. Την άποψή μου, όντω γνωρίζουμε ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα, θα γίνει ψηφοφορία, ακόμη πιστεύουμε ότι δεν είναι ο σωστό τρόπο τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Υπάρχουν και άλλοι του τομεί του οποίου θα πρέπει να δούμε πώ μπορέσουμε να. Ε, ε, και για, με λειτουργικά μέτρα και με, στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, πώς μπορούμε να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις για το περιβάλλον και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έγινε λάθος. Και το καλύτερο θα είναι να το αναγνωρίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε λάθη κάνουμε και να προχωρήσουμε. Διαφορετικά, εάν προσπαθούμε να επεκτείνουμε τα αυτό το οποίο είχε καταρχάς γίνει στον τομέα αυτό και μόνο, νομίζω ότι πάλι λάθος κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά τον ΙΚΑΟ, κατά ό,τι καταλαβαίνω, η συνέλευση του ΙΚΑΟ δεν ήταν πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Δεν είμαι απεσιόδοξη, αλλά δεν είμαι και αισιόδοξη. Δεν νομίζω ότι θα μας ε, δώσει την απάντηση ο ΙΚΑΟ. Τελικό ερώτημα είναι το εξή λοιπόν. Από την ΙΣΙΑ προς την Επιτροπή. Σε ένα χρόνο, όταν ακόμη και ο ΙΚΑΟ, πράγμα το οποίο δεν θα συμβεί, θα πρέπει να έχει βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, δεδομένου ότι ο ΙΚΑΟ δεν έχει την κυβέρνηση που επιτρέπει να μας πει τα κάνουμε, τι θα γίνει όταν κάποιες χώρες δεν θα έχουν συμμορφωθεί. Αυτό μπορεί να το κάνουν ε, οι ΙΠΑ, διότι η σχετική νομοθεσία τους το επιτρέπει. Τι θα συμβεί λοιπόν στο τέλος του έτους, όταν κι άλλες χώρες δεν θα συμμορφωθούν με το όλο θέμα αυτό. Κύριος Γκάλ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο μετά από αυτά που είπε και η κυρία Τζάκη Φώστερ. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπατε, κυρία Φώστερ. Και εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στις αεροπορικές εταιρείε. Αφενός ε, να έχουν αυτές τις επιβαρύνσεις, να διατηρήσουν αυτές τις επιβαρύνσεις και να πιέζονται παράλληλα από τον αραβικό κόσμο ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και να διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου μονομερός μόνο ισχύουν αυτά τα μέτρα σήμερα. Αυτό δεν είναι επωφελές. Και γι' αυτό καλό και τον Επίτροπο Χίντεγκαρτ να υπάρξει αναστολή των μέτρων αυτών μέχρι ότου βρούμε μια καθολική παγκόσμια λύση για το ETS. Για να μην βαρύνονται υπερβολικά μόνο κάποιοι από τους φορείς της αγοράς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να γραφεί στα πρακτικά ότι συμφωνώ απολύτω με του και πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να πω το εξή. Αν η κύρια ιδέα είναι να κάνουμε κάτι για να μην θεωρηθούμε ε, γελοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς θα κάνουμε ότι χειρότερο. Θα πρέπει να υπάρξει παγκόσμια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Σπέρκερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ εν συντομία να πω ότι θεωρώ Πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να αποφύγουμε τις τρευλώσεις του ανταγωνισμού εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιριών. Νομίζω ότι αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε να αναστείλουμε την εφαρμογή του συστήματος μέχρι ότου βρεθεί μια καθολική παγκόσμια λύση. Ιδάλλως θα είναι δραματική η κατάσταση για την ε, αεροπορία μας στην Ευρώπη. Υποστηρίζω λοιπόν αυτά που προτείνει ο κ. Ματιέ και αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Ευχαριστώ. Thank you. For myself, before I bring in... Πριν ε, να μιλήσει η Γενική Διεύθυνση από την Κομισιόν που είναι υπεύθυνη θα πω το εξή. Στην έκθεση του ο Ματιό Γκρός ανέφερε ότι θα πρέπει η γνωμοδότηση αυτή να όποια και να είναι η απόψή μα, να πάει στην Επιτροπή Ένβη. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια ιδιάζουσα κατάσταση υπάρχει σύγχυση. Εν πάση περιπτώσει, πρώτα απ' όλα εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε το ματιό Γκρός και την έκθεση που κατέθεσε. Δεύτερη παρατήρηση που αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο πολλά μέλη είπαν. Και θα ήθελα η Γενική Διάθεση για την Κλιματική Αλλαγή να απαντήσει ε, σε κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν. Μας απασχολεί στην Επιτροπή αυτή τι θα συμβεί εάν στην, με, δεν υπάρξει συμφωνία μετά τη Γενική Συνέλευση του ΙΚΑΟ. Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Και ξέρουμε ότι ο ΙΚΑΟ είναι ένας οργανισμός στον οποίο δύσκολα λαμβάνονται τέτοιου είδους ε, αποφάσεις και συμφωνίες, κυρίως για ένα τέτοιο θέμα. Και αν σταματήσει ο χρόνος, όπως λέγεται, και αρχίσει να γίνεται πόλεμος με τις εκπομπές και τα δικαιώματα, δεν ξέρω τι θα γίνει. περιπτώσει, πιστεύω ότι εμείς μπορούμε να πούμε καλόψε ότι θα θέλαμε να υπάρχει παγκόσμια συμφωνία. Αυτό είναι το κλειδί. Αλλά πιστεύω ότι με αυτό το θέμα πραγματικά θα μπούμε σε μεγάλο πρόβλημα εάν προχωρήσουμε έτσι όπως προβλέπετε. Και υπάρχει το θέμα των ε, στρεβλώσεων που θα δημιουργηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι πιστεύω ότι εμείς μπορούμε να το χειριστούμε το όλο θέμα των ETS, αλλά τι γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, συμφωνώ με τον Μάικρο ότι πρέπει να έχουμε μια εναλλακτική λύση και διαφωνώ με αυτό το οποίο λέγεται δεν θα είναι ενδεχομένω η απάντηση, η εναλλακτική λύση, το σχέδιο Β. Τώρα, τι θα γίνει αν και όλα αυτά τα σενάρια. Ίσως σας φαίνονται όλα απεσιόδοξα αυτά, Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε απεσιόδοξοι τα τελευταία χρόνια, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει εάν εφαρμοστεί το άλλο σενάριο και τι θα γίνει. Και πώς θα ενεργήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Αν δεν υπάρξει παγκόσμια συμφωνία. Δεν υπάρχει παγκόσμια συμφωνία και όταν αρχίσουμε εμείς να εφαρμόζουμε αυτό το σύστημα το ETS για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών, τι θα κάνουμε όταν θα ξαναβρεθούμε στην ίδια θέση με την οποία είχαμε βρεθεί πριν ε, να σταματήσει να εφαρμόζεται η οδηγία και να λαμβάνονται διάφορα μέτρα αντιπερισπασμού από διάφορες τρίτες χώρες. Αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα χειριστούμε και να δούμε τι γίνεται από την άποψη κλιματικής αλλαγής. Όχι να δούμε τα πράγματα με την οπτική γωνία ότι θα υπάρξει συμφωνία. Δεδομένου ότι υπάρχουν ενδιασμοί και υπάρχουν σκεπτικιστέ όσον αφορά το θέμα αυτό. Η κυρία Ηλεάνα Μπάντα από την Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτούς που εξέφρασε την εκτίμησή τους για το πόσο γρήγορα έκανε την έκθεσή του ο κύριος Γκρός. Και να, να γνωρίσω ότι η προσπάθεια που έγινε ήταν εξαιρετική και ό,τι κάνατε ώστε να μπορέσετε όλοι ε, να συνεργαστείτε σωστά ώστε να έχουμε αυτή την προσέγγιση και πλήρη γνώση του θέματος. Όντως είμαστε σε μία κατάσταση κατά την οποία ενεργούμε με ασυνήθιστη ταχύτητα. Πρέπει να υπάρχει βούληση και πραγματισμός για να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς να συνεργαστούν. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Έχουν γίνει οι συνεδριάσεις από τις ομάδες εργασίας από το Συμβούλιο και τώρα η Επιτροπή έχει λάβει και τα κατάλληλα πρώτα βήματα. Θα ήθελα να κάνω βασικά τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, η Επιτροπή θέλει να υπάρχει για το θέμα αυτό της παρέκκλησης πλήρης διαφάνεια. Νομίζω ότι στην ε, διαδικασία συναπόφασης θα πρέπει να είναι όλοι απόφαση, αλλά θα πρέπει να γίνουν όλα με το σωστό τρόπο και έγκαιρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορεί μεταξύ των διεθνών ε, εταίρων μας, των ε, κρατών μελών και όλων των ενδιαφερμένων που απαιτούν διαφάνεια και θέλουμε να υπάρχει προς όλους και για τα πάντα διαφάνεια. Όσον αφορά τα διάφορα θέματα τα οποία έθεσαν, ότι θα πρέπει να είναι όλοι ε, στο ίδιο επίπεδο, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες του παιχνιδιού, ώστε να μην υπάρχουν ε, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, μιλούμε για μία παρέκκληση για ένα χρόνο, απλή εξαίρεση, όπως λέγει το άρθρο 16, που μας δίνει την πλήρη σαφήνεια χωρίς ε, να επηρεάζει το σύνολο της οδηγίας για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπής και μας επιτρέπει να λάβουμε μετά από την διακήρυξη που θα γίνει σε επίπεδο ΕΚΑΔΟ τα κατάλληλα μέτρα. Πρόκειται λοιπόν για ένα προσωρινό μέτρο. Άρα δεν νομίζουμε ότι θα επηρεαστούν πάρα πολύ οι ίσοι κανόνες για όλους. Εντός Ευρώπης οι φορείς εκμετάλλευσης που συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τις ε, ενδοευρωπαϊκές πτήσεις πρέπει ούτως ή άλλως να συμμορφώνονται με την ε, κοινοτική νομοθεσία και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και για τις αναφορές και για τις ε, ε παράδοση των δικαιωμάτων εκπομπών. Τώρα, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο, θα πρέπει στα πλαίσια των τριλόγων και στι υπηρεσίες της Επιτροπής να συζητήσουμε τι θα γίνει μετά στα πλαίσια τη εφαρμογή των ε, διαφόρων μηχανισμών και αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε πρώτα εσωτερικά. Τελικά, για τη διαδικασία στο ΙΚΑΟ θα πω το εξή. Είναι σαφέ ότι όλοι θέλουμε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Και όλα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν Σεπτέμβρη-Κτώμηση. Παρά όλα αυτά πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας, διότι αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει την δυναμική των διαπραγματεύσεων. Και βεβαίως η... για να μπορέσουμε να κάνουμε τις κατάλληλες ε, διαβουλεύσεις και να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι εταίροι των τρίτων χωρών, θα πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς για το τι θέλουμε και βεβαίως να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα υψηλού επίπεδου ώστε να προσθεθεί σε όλη την διεθνική διαδικασία του ΙΚΑΟ για τα μέτρα αυτά τα αγορακεντρικά να προσδώσει και την πολιτική διάσταση είναι κάτι το οποίο θα επιτρέψει να δούμε σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούμε ώστε να μπορέσει ένα παγκόσμιο μέτρο να εφαρμοστεί, να γίνουν συζητήσεις για τις ε, δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής αυτού του παγκοσμίου μέτρου και σε τρίτο επίπεδο θα γίνουν συζητήσεις και για άλλα θέματα και τεχνικά μέτρα και ε, σχέδια δράσης που θα είναι επωφελής για άλλους. Θέλουμε αυτό το πακέτο λύσεις να είναι επωφελής για όλους με την εφαρμογή του ETS στο μεταξύ διάστημα. Θα πρέπει να συμφωνηθεί το γενικό πλαίσιο δράσεως και πιστεύουμε ότι στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας του ΙΚΑΟ θα μπορέσουμε να έχουμε σωστές διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και θα μπορέσουμε το σύστημα ETS να το εφαρμόσουμε και προς όλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριος Γκρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο σε σχέση που, με αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσαμε για ένα πλαίσιο, σύμφωνη. Αν σε επίπεδο ΙΚΑΟ προκύψουν θετικές ενδείξεις, θα ήθελα να υποδείξω το εξή θα είναι προς το συμφέρον και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεργαστούμε πολύ καλά και να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με αποφάσεις ε, οι οποίες απλά θα κοινοποιηθούν στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο δείχνει πολύ ανοιχτό χαρακτήρα για συζήτηση και δίνει το περιθώριο εφαρμογή ε, για να ληφθούν οι απαραίτητε διατάξει, Αυτό θα πρέπει να τηρήσουμε σαν αρχή. Είναι πολύ σημαντική πτυχή αυτή. Κάτι άλλο τώρα. Και να απαντήσω ίσω στην ερώτηση του Brian Simpson έτσι. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν έχουμε καμία άλλη εναλλακτική λύση παρά να πούμε το εξή. Αν δεν σημειωθεί η επιτυχία θα εφαρμοστούν αυτά που ισχύουν ω ευρωπαϊκή νομοθεσία σήμερα. Γιατί αν ε, σήμερα ξεκινάμε να ζητούμε εναλλακτικές λύσεις, σχέδιο Β, αποδυναμώνουμε και την δική μας ε, θέση και την ε, θέση όσων ψάχνουν γενικά μια παγκόσμια λύση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις. Θα ήθελα επίσης να καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα σήμερα το οποίο χρονικά θα μας επιτρέψει να χορηγήσουμε την γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τις τροπολογίες 28 Ιανουαρίου, μεσημέρι 12 η ώρα. Ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας. Η Επιτροπή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα γίνει 26 νομίζουμε και στην Ολομέλεια του Απριλίου για να τηρήσουμε τις προθεσμίες. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να θυμάστε Προθεσμία για την υποβολή των απολογιών 28 Ιανουαρίου 12 η ώρα. Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική μεταφορών της Ένωσης. Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του κυρίου Μαρινέσκου. Έχετε το λόγο κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Το 2005 πρώτο είδαμε το θέμα αυτό με ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Κατόπιν το 2006 άλλαξαν τα πράγματα. Λήφθηκαν, έγιναν βήματα προς τον μπρος σε συμφωνίες με τρίτες χώρες για την δημιουργία μιας κοινή ζώνης άρματα με τις ε, γειτονικές χώρες της Ένωσης. Ωστόσο, έχουμε, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, την αύξηση, τη μεγάλη, η, μεγάλη, α, η μεγαλύτερη αύξηση των αερομεταφορών αυτή τη στιγμή γίνεται στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, κάτι που σχετίζεται και με την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες εκείνες που προχωρά με ταχύτερο βήμα από ό,τι στην Ευρώπη. Από πλευράς μου, <coughs> θα έλεγα ότι αν θέλουμε να υπάρξει εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ένωσης πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε τα εσωτερικά προβλήματα που διαθέτουμε για να ολοκληρώσουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Κατά την άποψή μου, εδώ έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Γίνονται βήματα, αλλά δεν είναι επαρκή. Η ιδέα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού περιλαμβάνει και χώρες που είναι γειτονικέ χώρες στην Ένωση. Όταν λοιπόν συζητούμε με άλλες χώρες το θέμα αυτό και, θέτουμε, και θέλουμε να θέσουμε προϋποθέσεις ε, διεθνών συμφωνιών, θα πρέπει οι προϋποθέσεις αυτές να τηρούνται πρώτα στο εσωτερικό της Ένωσης. πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να δοθεί μια εντολή στην Επιτροπή για να, συν, για να διαπραγματευτεί με τους ατουγικούς εταίρους μας σε τέτοιες μορφές ε, διαπραγματεύσεων όπως Κίνα και Ινδία. Να λάβουμε υπόψη τις, ε, τους περιορισμούς που επιβάλλονται αυτή τη στιγμή στις αεροπορικές εταιρείες και να λάβουμε υπόψη το θέμα του εσωτερικού ανταγωνισμού. Και τα τέλη, τα εθνικά τέλη καθώς και τα τέλη επιβατών. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μία έκθεση που θα ενισχύει την προσέγγιση για μία συνεκτική πολιτική αερομεταφορών που θα ενθαρρύνει την γενική ανάπτυξη της οικονομίας, την ευρύτερη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια, στην παρούσα στιγμή και να εξετάσουμε τις θετικέ επιπτώσεις των άμεσων εμπορικών, του άμεσου εμπορικού ωφέλους για τις αερομεταφορές και τα πλονεκτήματα για τους επιβάτες. Ο κ. Αλκαντράουρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς ε, κύριε Σιγητά για την εισαγωγή σας. Βρισκόμαστε στη φάση σε μιας πρώτης συνταλλαγής απόψεων. Ανυπομονώ λοιπόν να δω πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Δύο στοιχεία θα ήθελα ωστόσο να τονίσω. Καταρχάς πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση των συμφωνιών σε σχέση με τις ε, αερομεταφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών των τελευταίων ετών και θα πρέπει να κοιτάξουμε εις βάθος κατά πόσον οι συμφωνίες αυτές ε, τελικά έχουν αποβεί και προς όφελος δικό μας. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι κάπως ασαφές στην παρούσα φάση. Συνάψαμε συμφωνίες, επιτρέψαμε να εισέλθουν στην αγορά μας ξένες εταιρείε. αλλά μια συμφωνία μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχουν ίσοι όροι ουσιαστικά σε επίπεδο ε, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και το καθεξής. Όσον δεν υπάρχουν ίσοι όροι, είναι δύσκολο να υπάρχει και δίκαιος ανταγωνισμό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε έχει να κάνει με το ότι αντιλαμβανόμαστε σε κάποιες χώρες γίνονται δημόσιες επενδύσεις και μάλιστα πολύ υψηλές ε, σε εθνικούς αερομεταφορείς. Και έτσι γίνεται στρέβλωση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Και κάτι τελευταίο, και εδώ θα συμφωνήσω με τον εισηγητή, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι και σε εμά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί κανόνε και πολλά διαφορετικέ συνθήκε αν θέλετε, μεταξύ κρατών μελών, όπω για παράδειγμα στι κοινωνικέ συνθήκε. Νομίζω ότι σε έναν τομέα όπω είναι οι αερομεταφορέ, θα πρέπει να κινηθούμε σιγά-σιγά προ μία κατεύθυνση εναρμονισμένης ε, νομοθεσία. Οδεύουμε προ το δρόμο αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μα ακόμη. Ευχαριστώ. Mr. Κύριος Μπένιον. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την έκθεση. Είχαμε δει και την ενημέρωση της Επιτροπής ε, σχετικά για το τι έγινε και τι πρέπει να γίνει. Πιστεύουμε ότι αν η Ευρώπη θέλει να μείνει κόμβος μεταφορών στην Ευρώπη πρέπει να έχει μια εξαιρετικά ισχυρή εξωτερική πολιτική αερομεταφορών και άρα οι αποφάσεις ε, της Ένωσης πρέπει να είναι συνεκτικές και να σέβονται, να καταλαβαίνουν τη διεθνή πραγματικότητα. Γι' αυτό η αξιοπιστία της εξωτερικής ε, πολιτικής είναι απαραίτητη και στην, στο διεθνή, για να έχουμε μια ενιαία φωνή και στον διεθνή οργανισμό αερομεταφορών. Καλή ιδέα είναι να δουν ολόκληρη την αλυσίδα ε, αξιών της ευρωπαϊκής, ε, των ευρωπαϊκών αερομεταφορών. Υπήρξε μια ανακοίνωση πρόσφατα των αεροπορικών εταιριών που εξέφραζαν ανησυχίες για τους περιορισμούς που προτείνονταν για τα αντιδιαβρωτικά. Κάτι που θα δυσκόλευε τη συντήρηση των αεροσκαφών ε, στην Ένωση. Δηλαδή θα έπρεπε να φύγουν εκτό της Ένωσης, να τους περάσουν τα αντιδιαβρωτικά και να τα ξαναφέρουν πίσω. Και υπάρχουν μάλιστα και κάποιες υποχρεώσεις ε, ε, που πρέπει να τηρηθούν για να προσγειωθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Καταλαβαίνω ότι αυτή η ανακοίνωση ξεπερνά τα πλαίσια των ε, αεροδρομίων. Χρειάζεται να έχουμε καινοτόμε λύσει. Ξεκινήσαμε κάτι τέτοιο ήδη. Υπάρχει έλλειψη χωρητικότητα στο χήθρο, για παράδειγμα, σε κάποιε περιπτώσει, Δημιουργούνται δεύτερε δεύτερες ε, εναλλακτικές ε, δεύτερη εναλλακτική κόμβη Τώρα για τα διεθνή εμπορικά θέματα, συμφωνώ απόλυτα με τους δύο προηγούμενους ομιλητές, πρέπει να δούμε πώς έχουν οι συμφωνίες μας όχι μόνο με Κίνα και Ινδία αλλά και με Ήπα. Στις ΗΠΑ η αγορά παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν ε, εμπορικέ διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ. Ίσως αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα τη ημερήσια διάταξη. Αυτά ευχαριστώ και προσβλέπω σε μια καρποφόρα συνεργασία. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή αυτό το θέμα να τρέχει και σε μια περίοδο πριν το 2005 όταν είχαμε τη συζήτηση για τους ανοιχτούς ουρανούς με την Επίτροπο κυρία Παλάθιο. Θα το θυμάται ο Μπράιαν, δεν ήσουν ο πρόεδρος βέβαια, θα το θυμάσαι. Είναι ένα θέμα που είχε μείνει στην συζήτηση για πολύ καιρό και σωστά. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών έκανε μεγάλα βήματα έκτοτε, παρότι δεν ήταν εύκολο. Η πραγματικότητα είναι ότι χρειαζόμαστε καλές συμφωνίες ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρότι υπήρχαν κάποιε επιφυλάξεις ε, όταν εξετάζαμε το ενδεχόμενο να κλείσουμε αυτές τι ε, συμφωνίες σε διμερέ επίπεδο. Υπήρξε πρόοδο λοιπόν, ακόμα και με τις Ηνωμένες που είναι βέβαια μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. Προφανώ πρέπει να προχωρήσουμε. Υπάρχουν χώρε όπου χρειάζονται συμφωνίε. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν θα σας πω πώς να διαπραγματευτείτε, αλλά αυτό που όταν ε, συνάπτουμε τέτοιε συμφωνίες με τρίτε χώρες, δεν είναι δεδομένο ότι θα πετύχουμε πάντα αυτά που θέλουμε. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να έχουμε κάποια συμφωνία και μετά να, δηλαδή πρέπει να πετύχουμε μια συμφωνία και να προχωρήσουμε κατόπιν. Το άλλο θέμα που είναι όντως αύξηση των μεταφορών στην Ασία, την Αμερική, η, δυνατότητα, η μη δυνατότητα των ευρωπαϊκών ε, αεροπορικών μεταφορών να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Ε, όλη η συζήτηση για το τέταρτο διάδρομα προς γύρω στο για παράδειγμα, το δείχνει για να μπορέσουμε να, συγχω... να, να, να συνεχίσουμε είμαστε αγωνιστικοί πρέπει να ανανεωθούμε. Ω εισηγήτρια για τον, ε, τη διαχείριση εναέριων μεταφορών για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό θέλω να υπογραμμίσω ότι η ευθύνη είναι το... αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί έχουμε επιχειρήσεις που είναι παγκοσμίου επίπεδου που βρίσκουν, αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνε τους στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία όφηση προς σωστή κατεύθυνση. Κλείνω λέγοντας ότι κάποια πράγματα όπως το ETS δεν βοηθούν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να αυξήσουμε υπερβολικά την νομοθετική ρύθμιση των ευρωπαϊκών αερομεταφορών. Αλλιώ είναι παγκόσμιε εταιρείε οι εταιρείε αυτές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, επιβάλλουμε συνεχεί κανόνες. Όχι ότι δεν προστατεύουμε τον καταναλωτή, αλλά υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε το ανταγωνιστικό μας πλονέκτημα για τους λόγου που ανέφερα. Κλείνω. Το θέμα δεν είναι θέμα μεταφορών μόνο. Εδώ υπάρχει μια τεράστια αλυσίδα ε, που συνδέεται από τον τουρισμό μέχρι τα, τις, ε, ε, τη συντήρηση. Μην την ξεχνάμε αυτή τη διάσταση. Υποστήριζω λοιπόν ε, την πρόταση, προτείνω στην Επιτροπή να προχωρήσει με τον επικοδομητικό ρόλο που παίζει μέχρι τώρα, να λάβει υπόψη κάποια από τα σχόλια. Όχι γιατί είμαι απεσιόδοξη, αλλά γιατί ρεαλιστικά πρέπει να δούμε τον ανταγωνιστικό μας χώρο. Αν θες να χτίσει αεροδρόμιο στη Μέση Ανατολή την Ασία δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν είμαστε γαλοπούλες που ψηφίζουν να έρθουν τα Χριστούγεννα νωρίτερα. Δεν πρέπει να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να μην μπορούν να ανταγωνιστούν ή να μπορούν να ανταγωνίζονται σε ένα τελείως δυσάρεστο ε, πλαίσιο. Ο κ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει. Όπως είπε και ο συνάδελφος Σάιτ, πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω όμως ότι τα διάφορα θέματα τα οποία επεξεργαζόμαστε τα τελευταίους μήνες εδώ πέρα καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι για μας για Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρούμε μία λύση για μία ευρωπαϊκή προσέγγιση στα θέματα αυτά. Και η πρόκληση έγινε στο ότι στο επίπεδό μας ε, θέτουμε ποιοτικά κριτήρια τα οποία ισχύουν και στον οικονομικό και στον περιβαλλοντικό τομέα για τις εργασιακές συνθήκες, για τα τεχνικά πρότυπα και τελικά αναρωτιέμαι είμαστε σε θέση να πείσουμε για τα ποιοτικά μας αυτά πρότυπα και τους άλλους ή μήπως όχι. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο ανακύπτει και θα πρέπει να το συζητήσουμε στο θέμα, στον τομέα αυτό. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν θέλουμε την πιο φτηνή λύση, αλλά την πιο καλή λύση. Και η πιο καλή λύση θεωρώ ότι δεν είναι πάντα αυτό το οποίο επιλέγει η αγορά, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να πιστούμε για τους παράγοντες αυτές. Τελευταία σημαντική παρατήρηση λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε ε, να αντιλαμβανόμαστε ότι στην Ευρώπη όσο μιλάμε με 27 διαφορετικές ε, φωνές δεν θα πείσουμε τους άλλους. Αναφέρθηκε και το Open Sky. Μια μεγάλη χώρα όπως η Αμερική δεν συνάπτει ε, συμφωνία με την Ευρώπη αλλά με 27 κράτη-μέλη όπου κάποιες χώρες δίνουν περισσότερα προνόμια υποστηρίζουν το καμποτάζ, για παράδειγμα. Ενώ ξέρουμε ότι στην Αμερική δεν ε, μπορούν να εφαρμόσουν το καμποτάζ. Το γεγονός λοιπόν ότι μιλάμε με 27 διαφορετικές φωνές και αφήνουμε τα πράγματα αυτά στις εθνικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας αποδυναμώνει σε πολιτικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Και αυτό αποτελεί ένα μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε. Εγώ στη χώρα μου ιδιαίτερος τα είδα αυτά και στη συζήτηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, πώς διαπιστώσαμε μετά από αξιολόγηση της κατάστασης ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάμε με μία φωνή. Και αυτό που ζούμε στο FAPS, όπου βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ενιαία φωνή και δεν μπορούμε να πείσουμε τις άλλες χώρες, παρόλο που είναι σαφές τι πρέπει να γίνει από τεχνικής άποψης, καταδεικνύει ποια είναι η αδυναμία μας. Θα πρέπει λοιπόν να αντιλαχθούμε ποιες είναι οι δυνατές μας, ε, τα δυνατά μας σημεία και ποια είναι τα μας σημεία μας. Ευχαριστώ κύριε Γκρός. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Μαρινέσκου για την αρχική εισαγωγή. Αναφέρθηκε ότι αυτό ήταν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Τρει τομεί θέλω να υπογραμμίσω ω κομμάτι της ε, δική μα πολιτική. Πρώτον, το πώ δουλεύει η ΆΣΕ σε παγκόσμιο επίπεδο ως ε, κανονιστική αρχή και αρχή επιστοποίηση. Αυτό ανέκυψε και πάλι την περασμένη εβδομάδα μετά την ιστορία των 787 η FAA και η ASA συνεργάστηκαν και νομίζω θα ήταν χρήσιμο να το δούμε. Να δούμε το πώς ε, γίνεται αυτή η επικοινωνία της EASA με άλλες ρυθμιστικές αρχές όπως την FAA. Δεύτερο θέμα. Το, το έθιξε η κυρία Φώστερ. Ο ρόλος της Ένωσης στον ΆΙΚΑΟ. Το είπε και ο κύριος Μπενιόν, νομίζω. Μερικές φορές μπορεί να δημιουργεί αμηχανία στην ΑΙΚΑΟ είναι τα κράτη-μέλη, όχι τα, τα, η Ένωση. Θα ήταν χρήσιμο να δούμε πώς δουλεύει αυτό. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι σωστή ο όρος πρόβλημα, αλλά ποια είναι η σχέση της Ένωσης όταν γίνονται οι μάχες στο εσωτερικό του ΙΚΑΟ. Τρίτο θέμα, Ρωσία και σχέσεις με Ρωσία. Ιδίως για τα, δικαιο, τα δικαιώματα υπερπτήσεων. Στην Ένωση αγωνιζόμαστε εδώ και καιρό να κάνουμε τους Ρώσους να είναι λίγο πιο λογικοί στα θέματα δικαιωμάτων υπερπτήσεων. Υπήρξε και μια σχετική επιστολή σχετικά μια, ένας βασικός ωστόσο, μια βασική παράμετρος της εξωτερικής μας πολιτικής στο μέλλον είναι οι σχέσεις μας με την Ρωσική Ομοσπονδία. Και τούτο το βλέπω ως αντίστοιχα σημαντικό με τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Αυτή είναι η τρεις τομείς νομίζω που πρέπει να εξετάσουμε και να καλύψουμε. Ο κύριος Μπόλτιν, Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σα, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθώ να βρω με κάποιον να διαφωνήσω, αλλά δεν γίνεται. Συμφωνώ. Ξέρω ότι τα τελευταία δεκαετία συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκο για την εργασία που θα κάνει τι παρατηρήσει που ήθελα. Υπάρχει και η εκθέση του κυρίου Λικαντράη του 2005. Πολύ σωστή και πολύ σωστά επισημάνατε αρχίζοντας παρατηρήσεις πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, πόσο σημαντικό είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, τι γίνεται με τα εθνικά τέλη, του εθνικού όρου, με τα έργα υποδομής και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, πόσο ε, σημαντικός είναι και ο ρόλος σε αυτή την περίπτωση. Απλώς θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Στην Επιτροπή, όπως και εσείς, αρχίζουμε από το ότι θεωρούμε πόσο στρατηγικός είναι και θεμελιώδης για την ανάπτυξη και τις επικοινωνίες ο ρόλος των ε, αερομεταφορών. Υπάρχουν ε, προβλήματα, αλλά έχουμε τρεις από τις δέκα καλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Έχουμε πέντε ε, εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, έχουμε 3,5% ποσοστό στην, του ΑΕΠ Όντω υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολε στιγμές για την αεροπορία και σε αυτό το πλαίσιο εμεί ε, κάνουμε, κάναμε στι αρχέ του έτου αναθεώρηση του όρου συστήματο, ήρθαμε σε επαφή με τα κράτη-μέλη, με όλου του εταίρου για να μπορέσουμε να δούμε εάν όντω και να κάνουμε αποτίμηση τη πολιτική την οποία αρχίσαμε για την αεροπορία από το 2005 και μετά και να δούμε πώ θα ανταποκριθούμε στι μελλοντικέ προκλήσει. Τα τελευταία δέκα χρόνια νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιες ήταν οι επιτάξεις μας. Οι σπηλώνες, ε, ισχυρή νομική βάση και σημαντικές συμφωνίες με εταίρους κλειδιά, πολύ καλά αποτελέσματα, εξε... χάρη στον ε, συντονισμό τον οποίο είχαμε, ξέρουμε ότι έχουμε γίνει πάρα πολλές ε, διμερείς εμπορικές συμφωνίες με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ έχει αναγνωριστεί και έχει οριστεί ο χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Μεταφορέα. Συμφωνίες με τις γειτονικέ χώρες, με το Μαρόκο, με την Ιορδανία, την Μολδαβία, τη Γεωργία, τις Βαλκανικές χώρες και άλλες συμφωνίες οι οποίες διαπραγματεύονται οικονομικά ωφέλη από την πρώτη συμφωνία με τη Δυτικά Βαλκάνια 6 δις ευρώ από το 2006 έως το 2011, τρίτο πυλώνα, και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τις διάφορες συμφωνίες τις οποίες έχουμε με την ΕΠΑ, με τον Καναδά και τη Βραζιλία. Τώρα, πρόκειται για μια αποδοτική πολιτική η οποία λειτουργεί, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε υποστεί μεγάλο πλήγμα στην Ευρώπη, υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των αεροπορικών εταιριών και υπάρχει και το θέμα των ETS. Όντω, πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε γρήγορε μεταφορέ τη πολιτική για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι προκλήσει, για να μπορέσουμε να έχουμε μία ε, βιομηχανία πάρα πολύ ανταγωνιστική και σε θέση να ταξιδεύει άνω τον κόσμο. Επίσης, υπάρχει εθνικός κατακαιρματισμός των ευρωπαϊκών ετών. Υπάρχει έλλειψη ενότητας, λοιπόν, έλλειψη αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμφωνώ πλήρω με αυτό το οποίο είπε ο κ. Γκρός για το θέμα αυτό και κατανοώ και αυτά που είπατε και εσείς και η κυρία Φώστερ για το πόσο σημαντικό είναι το ΕΚΑ και πόσο σημαντικό είναι εμείς να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όμως δεν θα αλλάξουν βράχη πρόσφατα το μεσοπρόσφατα τα πράγματα αλλά τα μέτρα του μεσοπρόθεσμα και κυρίως ο συντονισμός, συντονισμός, ο συντονισμός μεταξύ ημών και των εταίρων μας είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ισχυρό μέτωπο ευρωπαϊκό σε επίπεδο ΕΚΑ. Τώρα, η ενοποιημένη θέση της Ευρώπης, όπως ξέρετε, από την κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζεται η Ρωσία, ε, τίθεται σε αμφίζηση. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση. Εκεί θα πρέπει όντως να μιλούμε όλοι με μια φωνή. Και τώρα έχει να αναγνωρίσει έχουν ευρύτατα τα κράτη-μέλη ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τη Ρωσία όντως μπορεί να δημιουργήσει δύσκολες κατάστασεις. Όσον αφορά τα θέματα επικοινωνίας, προσπαθούμε όλα αυτά τα θέματα να μην τα λύσουμε ε, στη θεωρία, αλλά με πρακτικά μέτρα και πολιτικές, ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεσοπρόθεσμες μετά στην αγορά, την παγίωση των ε, αεροπορικών μας εταιριών. Είναι σημαντικό να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες για όλους, υγιής ανταγωνισμός και λαμβάνοντας υπόψη και τους μελμούς της οδηγίας. Και τώρα επανέρχομαι στο πόσο σημαντικό είναι αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη βεβαίως είναι σαφές ότι εάν διαπραγματεύονται μόνα τους δεν μπορούν να προοδεύσουν τον ίδιο τρόπο και οι διάφορες ε, ε όπως ξέρετε ε, συμφωνίες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην νότητα της Ευρώπης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα επωφεληθεί πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, αν υπάρχει μια σωστή εξωτερική πολιτική στον τομέα αυτό, θα δοθούν νέε δυνατότητε στην βιομηχανία και θα μπορέσουμε να προστατευτούμε όλοι από την ε, προβλήματα του και τις τρευλώσεις σε θέματα του ανταγωνισμού. Ε, μας ε, ικανοποιούν τα πορίσματα του Συμβουλίου. Θα θέλαμε κάπου να είναι λίγο πιο αλλά νομίζω ότι πραγματικά γίνεται σωστός και επιδικομητικός διάλογος και θα θέλαμε να έχουμε και τη δική σας υποστήριξη, ώστε να έχουμε μία πάρα πολύ φιλόδοξη στη εξωτερική πολιτική στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μαρινέσκου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάνα δύο σχόλια μόνο θέλω να κάνω. Πιστεύω ότι τα σχόλια των συναδέλφων κατέστησαν σαφές ότι είναι πολύ πλοκό το θέμα και πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα κείμενο στο οποίο θα υπάρχουν συγκεκριμένες ιδέες για την πολιτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε τα πλαίσια τη εξωτερική πολιτική των αερομεταφορών. Θέλουμε η πολιτική αυτή για τα επόμενα χρόνια να είναι σωστή, ξέροντας ποιο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την η Ευρώπη να μιλάει με μία φωνή και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Η παρουσίαση της γνωμοδότησης θα γίνει 18-19 Μαρτίου στην συνάντηση Επιτροπής και θα έχουμε προσθεσμία κατάθεση τροπολογιών την 27 Μαρτίου και ψηφοφορία θα γίνει 22 και 23 Μαΐου. Η παρουσίαση Λοιπόν, τη έκθεση, επαναλαμβάνω, 18-19 Μαρτίου τον κύριο Μαρινέσκου. Προθεσμή κατάσταση τροπολογιών 27 Μαρτίου. Εξέταση των τροπολογιών 22 και 23 Απριλίου στη συνεδρίασή μας και ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στην συνεδρία της 7 Μαΐου. Εντάξει. Ε, καλώς, ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξη είναι η στρατηγική για μια υπηρεσία τηλεδιοδίων και ένα σύστημα αυτοκόλλητων σημάτων για τα ελαφρά οχήματα για ταχύ στην Ευρώπη. Είναι εδώ, Τζιμ. Είσαι εδώ. Τζιμ, το ξέρω. Θα σε πείραζε να περιμένουμε δέκα λεφτά γιατί δεν είναι κανένας από τους σκιώδεις ηγητής παρόντες στην αίθουσα. Δέκα λεπτά λοιπόν. Διαλυματάκι για καφέ, λένε και οι Αμερικανοί. Κυρία Higgins, Jimmy. Συμφωνείς? Οκ. Έχει καλώς. Δέκα λεπτά λοιπόν διάλειμμα.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 ξεκινήσουμε λοιπόν και πάλι. Ε, συνάδελφοι, μιλάμε για τη στρατηγική για μια υπηρεσία τηλεδιοδίων και ένα σύστημα αυτοκόλλητων σημάτων. Τζιμ, ευχαριστώ πρόεδρα για να σας εξηγήσω πού βρισκόμαστε και από πού προερχόμαστε. Εδώ και κάποιο καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να ελευθερώσει την διασυνοριακή ε, κυκλοφορία. Οι πρώτες απόπειρες ε, στο θέμα αυτό είχαν να κάνουν να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε ε, στρέβλωση της ιστορικής αγοράς λόγω σχετικών τελών. Και άρα, επειδή οι υποδομές της Ευρώπης ε, πλέον ε, έχουν παλιώσει και πρέπει να ανανεωθούν, αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την τις υποδομές χωρίς να στρεβλώσουμε μελλοντικά την ιστορική αγορά. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η αρχή του ρηπαίνων πληρώνει θα τηρηθεί και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ε, για να εφαρμοστεί ε, ένα σύστημα ηλεκτρονικών τηλεδιοδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, καταρτήσει δύο ανακοινώσει, μία για τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν τέλη για τι υποδομές των δρόμων σε ελαφριά οχήματα και άλλο ένα για το ηλεκτρονικό σύστημα επιβολής τελεδιοδίων. Τα δύο ε, έγγραφα ε, είναι σχετικά, αποτελούν σχετικά ζητήματα. Η διαδικασία είναι αργή και θα πρέπει να πούμε ότι τα αποτελέσματα συνολικά ήταν απογοητευτικά, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ίσως να είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή να καταρτήσει πιο δυνατή νομοθεσία για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα η e e σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Σύστημα Τηλεδιοδίων φαίνεται ότι το βασικό θέμα είναι κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, διατίθενται να ε, συσκεφτούν, να διαβουλευτούν για να εξυπηρετήσουν τον χρήστη των ε, δρόμων. Άρα το θέμα είναι πολιτικό και εμπορικό, όχι τεχνολογικό. Ως εισηγητής πιστεύω ότι η δυνατότητα να υπάρχει μία μονάδα η οποία θα χρησιμοποιείται σε όλους τους δρόμους για διόδια είναι δυνατόν. Αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κανένα τρόπο να αναγκάσουμε του εμπλεκομένου φορεί να το πετύχουν αυτό. Μία άλλη δυνατότητα είναι να υπάρχει διόδια χωρί ε, εμπόδια. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την εξετάσει επαρκώ αυτή τη δυνατότητα. Συστήνουμε να ληφθούν παρτερό μέτρα για να εξετάσουμε τη χρήση αυτού του συστήματο. ενδεχομένω σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ σε Ευρωπαϊκή, ως ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε μια ρεαλιστική λύση καταρχάς. Άκουσα τις ανησυχίες των εμπλεκόμενων φορέων σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα. Ωστόσο, η εισαγωγή ενός ενιαίου συστήματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολύνει τη ταξίδια. Η δημιουργία ενός σωστού συστήματος ή ETS θα πετύχει την άνεση των μεταφορών και θα μειώσει και το κόστος. Η υπερτέρω ανάπτυξη του ETS θα γλιτώσει και χρόνο και κόστος από τις σχετικές εταιρείες. Θα υπάρχει μόνο ένας λογαριασμός, γιατί οι οικονομίες κλίμακας δεν ε, θα ε, ωφελήσουν το σύστημα. Επίσης θα συνεχίσει να ισχύει η αρχή του ορυπένων πληρώνει. Ως θα πρέπει να συναντηθώ και με κάποιους ε, άλλους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά θα πρέπει να ε, λαμβάνω υπόψη και διάφορες πτυχές που θα αφορά αυτή η έκθεση και σε αυτή τη φάση ανυπομονώ να λάβω και προτάσεις από άλλους ευρωβουλευτές αλλά να ακούσω και την άποψη των σκιωδών. Τα κράτη-μέλη που θέλουν ένα σύστημα βάση χρόνου θα πρέπει να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν αυτό το σύστημα, αλλά οι τιμές που θα ε, επιβάλλουν ως τέλη θα πρέπει να είναι αναλογικές ε, ημερήσιες, ε, μηνιές, εβδομαδιές, χρο, ετήσιες, ε, ετήσιες ε, ετήσια, ποσά και θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αυτοκόλλητων. Το, για παράδειγμα, το αυτοκόλλητο για μία εβδομάδα θα πρέπει, για ένα μήνα θα πρέπει να είναι ε, ανώτατο όριο αντίστοιχο τέσσερις φορές ε, το εβδομαδιαίο. Σε ό,τι αφορά τα αυτοκόλλητα, τα κρατημέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέτοια τέλη, να χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση για τις υποδομές τους. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο σαφείς οδηγίες, προκειμένου να μπορούν να χρεώνουν προοράτα, με μικρή διοικητική επιβάρυνση. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πάει αρκετά μακριά στις προτάσεις της. Σύμφωνο με την άποψη ότι μια τέτοια βινιέτα θα πρέπει να είναι απλή στη χρήση για τους ε, οδηγούς και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εστιαστούν σε μία βινιέτα, σε ένα σύστημα αυτοκόλλητων που θα είναι δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης κάνει κάποιες προτάσεις για τις κυρώσεις και για την εφαρμογή και σε ό,τι αφορά την δυνατότητα αγορά τέτοιων αυτοπόλητων από τους οδηγού Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ρυθμίσει και το θέμα των μελλοντικών ε, επιβολών χρέωσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με συντονισμένο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οδηγίε δεν λειτουργούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει αρκετά για να διασφαλίσει ότι το ETS θα καταστεί ένα ρεαλιστικό σύστημα το οποίο θα εφαρμοστεί. Ελπίζω ε, οι πάροχοι υπηρεσιών κάπως να συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα EETS, αλλά θεωρώ ότι αν το αφήσουμε σε αυτούς, στα χέρια αυτών, δεν πρόκειται να προκύψει τίποτα. Είναι μη ρεαλιστικό αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα θέλαμε να σταλθεί στις 5 Φεβρουαρίου για μετάφραση το σχέδιο της έκθεσης, 7 Μαρτίου να το συζητήσουμε. 20 Μαρτίου είμαι τρόπο... ημερομηνία καταληκτική για κατάθεση τροπολεπηγιών. 23 Απριλίου να την ψηφίσουμε εδώ στην ε, Επιτροπή και 2 Μαΐου να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Είναι κάπως φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, αλλά ελπίζω να είναι πραγματοποιήσιμο. Γιατί θα πρέπει να θέσουμε κάποιους στόχους και κάποιες ε, καταληκτικές ημερομηνίε. Αυτά λοιπόν προτείνω στην Επιτροπή μας σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κ. Αλκαντράουι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χιγίνση για την εισαγωγή του. Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά, γιατί τα πιο πολλά από αυτά που μου ανέφερε ουσιαστικά συνάδουν και με τις δικές μου απόψεις. Και ξέρω φυσικά ότι εστιαζόμαστε στις ε, ε, εμπορικές μεταφορές. Θα ήθελα όμως να συμπεριληφθεί και κάτι σε ό,τι αφορά τη μεταφορά ατόμων, γιατί βλέπουμε ότι πολλά κράτη-μέλη αναλογίζονται το πώς μπορούν να χρεώνουν και τα ιδιωτικά οχήματα μέσω αυτοκόλλητων, βινιέτων κτλ. Αλλά συχνά αντιμετωπίζουν το εξής πρόβλημα. Η Ευρώπη μέσω κανόνων ε, κατά της διακριτικής ε, μεταχείρισης δεν αφήνει τα κράτη-μέλη να αντισταθμίσουν αυτές τις επιβαρύνσεις ε, με κάποιες ελαφρύνσεις σε άλλους τομείς. Και θα πρέπει να κάνει μία εις βάθος ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως να ε, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά τελικά δυσχεραίνουν την εφαρμογή νέων ε, ε, συστημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι χρησιμοποιούνται νέα συστήματα και είναι απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να οριστούν τεχνικά πρότυπα να διασφαλιστεί και η λειτουργικότητα, Γιατί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε να συμβεί στις μεταφορές ε, ατόμων αυτά που συμβαίνουν στις μεταφορές εμπορευμάτων. Γιατί συμφωνούμε νομίζω ότι τα αποτελέσματα του ETS ε, είναι απογοητευτικά και τα πιο πολλά κράτη-μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει τέτοια σύστημα τηλεδιοδίων τα έχουν πράξει αυτό χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τη μελλοντική ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της υπηρεσίας και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο αποφασιστικά προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα τα οποία χάνονται και πολύ αποδοτικότητα η οποία χάνεται. Και νομίζω ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Mr. Klins. Κύριος Κλίντς, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ με την θέση του κυρίου Higgins, του εισηγητή. Ως ε, κανονικοί πολίτες όταν μετακινούμαστε στην Ευρώπη, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήματα και σε πολλές περιπτώσεις θεωρούμε ότι είναι άδικη η μεταχείρισή μας. Ο σκοπός μας λοιπόν θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη να υπάρχει ένα καθολικό σύστημα ενιαίο, όπως είπε και ο εισηγητής, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα προοράτα για μία μέρα, για ένα μήνα, για ένα έτος να πληρώνει κανεί για να χρησιμοποιεί του δρόμους. Αυτό δεν ισχύει στην παρούσα φάση. Υπάρχουν πάρα πολλέ μεγάλες διαφορές και η δική μου χώρα δεν έχει κανένα σύστημα ουσιαστικά, ούτε το σύστημα αυτοκόλλητων, ούτε σύστημα τηλεδιοδίων, ούτε σκοπεύει να εισαγάγει ένα τέτοιο σύστημα. Και αυτό οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση λέει ότι είναι μεγάλη η επιβάρυνση ιδιαίτερα των ιδιωτικών οχημάτων. Υπάρχει και ένας σχετικός φόρος για τα οχήματα, υπάρχει φόρος στη βενζίνη και όλα αυτά αρκούν. Εγώ θεωρώ ότι στο πρόβλημα των διοδίων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το σύστημα διαφορετικής φορολόγησης των οχημάτων όχι μόνο τον φόρο της βενζίνης, τον φόρο των οχημάτων. Και μια χώρα η οποία εισαγάγει ένα σύστημα αυτοκόλλητων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει απαλλαγές και ελαφρύνσεις στο σύστημα φορολόγησης οχημάτων. Διαπιστώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε πετύχει την πρόοδο που θα θέλαμε. Αυτό το διαπιστώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θέμα είναι κατά πόσον θα μας βοηθήσει μια οδηγία ή κατά πόσον θα πρέπει να ακολουθήσουμε ε, τον οδό του κανονισμού. Επίσης, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα των διαφορετικών συστημάτων. Τρίτον, δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των μεταξύ των ε, χρηστών του δρόμου. Δηλαδή δεν ήταν να πούμε ότι α, διαφορετικά πράγματα ισχύουν για τον Αλαταπό, διαφορετικά ισχύουν για τον Ιμεδαπό, ε, χρήστη των οχημάτων, των δρόμων. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει συγκρισιμότητα, να ξέρουμε από τι αποτελείται το διόδιο το οποίο καλεί, καλείται κάποιος να πληρώσει, να υπάρχει το προράτα δηλαδή, συν κάποιο περιορισμένο διοικητικό κόστος. Πέμπτον, συμφωνώ τα κράτη-μέλη να καθορίζουν τα ίδια το ύψος των διοδίων. Γιατί είναι τόσο διαφορετικές οι συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη που δεν είναι δυνατόν μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια διαδικασία ανάπτυξης των υποδομών της, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, να επιβάλλει τα ίδια διόδια όπως η Ιταλία, η Γαλλία και το καθεξής. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, σαφώς σε ό,τι αφορά τώρα τα, τα φορτηγά. Νομίζω ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι όντω σε όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιηθεί η πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Ένα σύστημα υψηλής τεχνολογικής ε, προδιαγραφής που θα επιστρέψει στους ε, οδηγούς των φορτηγών χωρίς επιπλέον γραφειοκριτικό κόστος ε, να μετακινούνται σε όλη την Ευρώπη. Διασυνοριακά αυτό υπάρχει σήμερα ήδη. Θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά οχήματα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση να απλοποιηθεί το σύστημα αυτοκόλλητων. Να μπορεί να υπάρχει για παράδειγμα δυνατότητα αγορά στο διαδίκτυο, online. Μόνος του να το αγοράζει ο οδηγός. Όπως το βγάζει για παράδειγμα ο χρήστης αεροπορικής εταιρεία στο ίντερνετ του boarding card την κάρτα επιβίβασή του. Ξέρω, για παράδειγμα, εγώ περνάω από τη Γαλλία, την Ελβετία και τη Γαλλία και την Ιταλία και να ξέρω ότι μπορώ να βγάλω online το, το αυτοκολλητό μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Higgins διότι με μεγάλο θάρρος αντιμετώπισε το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ φιλόδοξο στόχο. Θέλουμε το σύστημα να λειτουργήσει σύντομα. Για τα φορτηγά δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη ένα ευρωπαϊκό σύστημα αυτοκόλλητο, ακόμη και στη χώρα μου. Τι σημαίνει αυτό, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το κατορθώσουν το σύστημα αυτό και η Ευρώπη παρομοίω. Μπορεί οι διάφορες χώρες να αποφασίσουν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα ή όχι, αλλά θα ήθελα να πω ότι είναι διαφορετικές οι επιθυμίε που εκφράζονται από κάθε χώρα και αν θέλουμε να έχουμε για τα ΙΟΤΑΧΗ ένα ενοποιημένο σύστημα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει και από πολιτική πλευρά η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμη και για τα φορτηγά. τα έσοδα από τους έμεσους φόρους στα καύση πρέπει να πω ότι δεν πηγαίνουν για έργα υποδομής το δικού δικτύου. Πράγμα που σημαίνει ότι τέτοιου είδους τέλη, ενδεχομένως οι φόροι, θα βελτιώσουν το δικό σύστημα. Αλλά υπάρχουν όντω μεγάλε διαφορέ όπω μεταξύ Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία. Και αν χρησιμοποιήσουμε για όλη την Ευρώπη αυτό το ενοποιημένο σύστημα, δεν ξέρω πώς θα το κατορθώσουμε. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ε, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στο δικό μας επίπεδο για το πόσο καλά πληρώνουμε τους ε, βοηθούς μας. Καταλαβαίνετε ότι στην Δανία Φερρυπίνο ο βοηθός ε, μπορεί να παίρνει 10-11 φορές ε, περισσότερα χρήματα από ότι ο βοηθός ενός Βουλγαρού. Αν μπορούσαμε να τα ενοποιήσουμε όλα, κάτι θα κάναμε, αλλά νομίζω ότι λάθος προτεραιότητες έχουμε θέσει. Ο κύριος... Ευχαριστώ τον κύριο Higgins που ανέλαβε το θέμα αυτό και για τις παρατηρήσεις που έκανε. Τον ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, η Επιτροπή πίστεψε ότι το θέμα αυτό ίσως θα ήταν εύκολο να εφαρμοστεί δεδομένου ότι υπάρχει πρόοδος της τεχνολογίας, αλλά η πολιτική κατάσταση είναι διαφορετική. Δεύτερη παρατήρηση. Ήδη τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις ε, ε, προκλήσεις που τίθενται και σε όλα τα ερωτήματα από πολιτικής, τεχνικής και τεχνολογικής. Γιατί με το σύστημα του GPS μπορούμε να καθορίσουμε κάποια θέματα σε σχέση με την ζώνη, με το τι είναι πληρωτέο, με το που ε, βρίσκεται κανείς. Υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα, χωρίς να έχουμε... έχοντας διαφοροποιημένα κόσμο και κάθε χώρα. Δύο ερωτήσεις θέτω, διότι τελικά Νομίζω ότι με το GPS θα καταλήξουμε στην εφαρμογή ενός πλήρως ψηφιωμένου συστήματος. Τι γίνεται με το θέμα του απορρίτου των δεδομένων και την δυνατότητα που υπάρχει για να τις χρησιμοποιήσει κανείς όπου θέλει. Για την εχνηλασιμότητα των μετακινήσεων, για τον εντοπισμό κάποιων και για την χρησιμοποίηση αυτού του συστήματος για άλλους λαούς. Δηλαδή ξέρουμε ότι αυτό το σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ενηχθευτούν διάφορες παραβάσεις του ΚΟΚ. Αυτό το σύστημα όταν έχει το GPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Πώς θα προστατεύονται οι χρήστες κατά οποιασδήποτε κατάχρησης ε, δεύτερον όταν έχουμε να κάνουμε με διόδια χωρίς ε, ε, μπάρα και να μην σταματάει κανείς, όπως γίνεται όταν έχει ε, κανείς την κατάλληλη ψηφιακή κάρτα, πώς μπορεί να ενημερωθεί ο χρήστης για την τιμή την οποία θα πρέπει να καταβάλει για το τμήμα αυτό το οποίο θα διανύσει χωρίς να σταματήσει. Να ξέρει εκ των προτέρων δηλαδή αν πάρει αυτό το αυτό τον αυτοκινητόδρομο, χωρίς να χρειαστεί να σταματήσει και να ξέρει πόσα θα πληρώσει, πώς μπορεί να ενημερωθεί έγκαιρα. Διότι δεν ε, μπορεί ο χρήστης όταν αλλάζουν οι τιμές ή όταν είναι διαφορετικές ή όταν δεν ξέρει ε, να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Δύο θέματα λοιπόν. Το απόρριτο και εκ των προτέρων ενημέρωση του χρήστη για το πόσο θα του κοστίσει να πάρει αυτό το κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου, διότι ενδεχομένω θα περάσει από ένα άλλο δευτερεύοντο δρόμο. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάλα Σέντερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τα σχετικά προς τον κύριο Χίνγκ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το όλο θέμα, το οποίο από Θεωρητική ίσως πλευράς όσον αφορά την, ε, τα τέλη αυτά και τα τηλεδιόδια και το σύστημα αυτοκόλλητων ε, σημάτων και σημαντικών και είπαμε ότι θα πρέπει να βασιστούμε στη νομική βάση. Βεβαίως θα πρέπει όλο και περισσότερο το θέμα αυτό να το χειριστούν τα κράτη-μέλη ε, και ο Γιάννης μιλάει όχι μόνο για γεωταχή αλλά και για τα μοτοποδήλατα, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιους. Τώρα, όσον αφορά το θεωρητικό μέλος, του ορισμούς, πιστεύω ότι η αρχή ο χρήστης πληρώνει και ο ρηπαίνων πληρώνει, πρόκειται για έννοιες οι οποίες όλο και περισσότερο περνάνε, αλλά στην εποχή αυτή που διερχόμαστε με την κρίση, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε το σύστημα αυτό όχι μόνο όσον αφορά το τι θα μας προφέρει τώρα, αλλά όπως κάνουν και οι Αμερικανοί, τι είδου ειδήσεις πρέπει να γίνουν και τι θα μας αποφέρουν. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε στη συζήτηση αυτή να τα θέσουμε. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Δεν ε, θα πρέπει τελικά με τέτοιου είδους μέτρα φτάσουμε στο άλλο άκρο. Να περιορίσουμε την ελεύθερη διακίνηση και να επιβάλλουμε ε, οικονομικά βάρη μεγάλη. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε και ποια χρησιμότητα. Τώρα είδαμε για να δώσω ένα παράδειγμα το θέμα των ε, ταχογράφων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε κάτι χωρίς μεγάλο διοικητικό άχθος και να δούμε το ε, κόστος. Είπε ο ότι τα μηνιαία τέλη θα πρέπει να είναι τέσσερις φορές τα εβδομαδιαία ή να δούμε πώς θα καθορίσουμε τις τιμές. Νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, ε, να δούμε τι γίνεται στην ε, Γερμανία, όπως είπε ο κύριος Ρικέ, ώστε να μην... Ε, ε, και όπως είπε και ο κύριος Ρικέ, να δούμε τι γίνεται με την εκ των προτέρων ενημέρωση των χρηστών για να δουν αν ως εναλλακτική λύση δεν θα ήθελαν να πληρώσουν αλλά να πάρουν ένα δευτερεύοντα δρόμο να φτάσουν εκεί που φτάνουν. Θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα δούμε. Και βεβαίως να δούμε κατά πόσο το σύστημα αυτό δεν αφορά μόνο τα δελταχή αλλά και τα ΙΟΤΑΧΗ. Τώρα, για την ε, ευρωπαϊκή κινητικότητα για και κυρίως για τις περιφερειακές χώρες της Ευρώπης. Να κάνουμε κάτι το οποίο σημαίνει συμπληρωματικό κόστος, δεν νομίζω ότι θα είναι και καλό αδεχθό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε. Και να δούμε πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και οι νέες οικογένειες που δεν έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, που ζουν ε, πολύ συχνά εκτός κέντρου της πόλης, αν πρέπει για να ξαναγυρίσουν, για να πάνε στο κέντρο της πόλης, να πάνε στη δουλειά τους, να ε, υποστούν ε, μεγαλύτερο κόστος, τι κάνουμε. Ο κύριος Καντσάν, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Χινής για την παρουσίασή του αυτή. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι πρέπει να απλοποιήσουμε οπωσδήποτε την ζωή του χρήστη, του πολίτη, του καταναλωτή. Εγώ ξεκινώ από ένα δεδομένο. Μιλούμε για μια οδηγία του 2004, πριν από 10 χρόνια δηλαδή. Αυτά τα χρόνια, μετά από τα χρόνια αυτά εξελίχθηκε η τεχνολογία, άρα η αφετηρία είναι ήδη λάθος. Δεύτερον, οι διαχειριστές των δρόμων δεν είναι πλέον ένας ανακράτος, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ τα λεγόμενα ΣΒΙΤ, η κοινή διαχείριση δηλαδή μεταξύ ιδιωτών δημοσίου. Η διαχείριση, άρα κάθε φορέας έχει δικά του έσοδα, δικά, δικές του εισόδους, δικές του εξόδους, Και αυτό διαπιστώθηκε όταν η εταιρεία του έργου παρουσιάζει στον δημόσιο φορέα την πρότασή της. Με αυτά τα δεδομένα, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή του πολίτη και να την καταστήσουμε απλούστερη, πιστεύω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Είτε να πάμε προς την κατεύθυνση των διοδίων χωρίς ε, μπάρες, υπάρχουν τα τεχνολογικά εργαλεία για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, ή να ενοποιήσουμε τις κατηγορίες διοδίων μεταξύ ποιου χρησιμοποιεί, ποιου ρηπαίνει, άλλα επιχειρία, άλλες παραμέτρους αν θέλουμε, αλλά να ενοποιήσουμε στο ίδιο διόδιο τους διάφορους τρόπους. Πιστεύω ότι με αυτές τις δύο με αυτά τα δύο βασικά στοιχεία πρέπει πραγματικά να επιδιώξουμε να δώσουμε απάντηση στο ζήτημα αυτό που έχει γίνει εξαιρετικά επίγον και όλοι περιμένουμε να δώσει η Ευρώπη μια σαφή απάντηση. Και από την οπτική των διαφόρων δομών και εναλλακτικών στα κράτη-μέλη και από την οπτική των, ε, της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό νομίζω είναι το επίγον. Αυτά είναι τα επίγοντα. Κύριος Μπένιον. Θεωρητικά υποστηρίζω τα διόδια εδώ και πολλά χρόνια, αλλά θεωρητικά αποκλειστικά. Θα μας πούν οι οικονομολόγοι και συνεχίζουν να μας το λένε συνεχώς ότι η τιμολόγηση της χρήσης των δρόμων είναι ο μόνος ορθολογικός τρόπος φορολόγησης ε, της χρήσης τους. Ε, ορθολογικά είναι σωστό. Αν ωστόσο το δείτε από την οπτική γωνία του ιδιοκτήτη του Ιωταχή, είναι πολιτικό δηλητήριο. Και να ήταν εγγυημένο ότι θα ήταν ουδέτερο φορολογικά θα υπήρχε μια απόλυτη εξαγρίωση των γεωταχίδων. Αν λοιπόν προχωρήσουμε σε κάτι μόνο για τα φωτιγά τα εμπορικά οχήματα μπορούμε. Κρίμα, αλλά μπορεί να είναι καλύτερο από ότι φερειπίν ε, τα τέλη κυκλοφορίας ή ε, η φορολόγηση των καυσίμων, αλλά υπάρχει τέτοια, τέτοια αντίδραση από τον κόσμο που δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή σε, οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πέραν των ε, φορτηγών. Γι' αυτό είναι θαραλέα η προσέγγιση του Τζιμ να προχωρήσει με το ζήτημα αυτό. Φοβόντουσαν όλοι νομίζω να βάλουν το όνομά τους δίπλα στην έκθεση. Βέβαια, αξίζει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για τα εμπορικά οχήματα όλο και περισσότερο αυξάνει την κυκλοφορία τους, ε, η διαχείρισή τους είναι περίπλοκη, υπάρχει... Σε κάποια κράτη-μέλη είναι πεπισμένοι ότι οι φωτιγατζίδες από άλλο κράτος μέλος έχουν μεγάλα πλονεκτήματα. Αξίζει λοιπόν να δούμε την προσέγγιση αυτή. Μέχρι εκεί θα σταματούσα τώρα. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι καλή ιδέα, αλλά πολιτικά δεν στέκει. Και συμφωνώ και με τον κύριο Ρικέ. Δουλέψαμε πολύ για το θέμα αυτό. Και στο κόμμα μου είχαμε προτείνει πολιτικές, οι οποίες κατόπιν είχαμε κάνει προτάσεις πολιτικών που εγκαταλείφθηκαν σε γαλήνια και χωρίς φασαρία όταν ετοιμάστηκε το μανιφέστο μας. Διότι ήταν, αυτό ήταν το βασικό θέμα ότι τα στοιχεία που θα συλλέγονταν δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιούσαν. Θέλουμε εγγυήσει γι' αυτό και ακόμα δεν είμαι πεπισμένο ότι μπορούμε να δώσουμε τι σωστέ εγγυήσει, την προστασία για την αποφυγή παράνομη χρήση των στοιχείων. Με εξότου υπάρξει εξασφάλιση γι' αυτό, θα υπάρχει και δεύτερο πρόβλημα. Αλλά προχωρήστε. Δείτε, φτιάξτε καμία πρόταση να δούμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω όμω ότι θα πρέπει να προσδοκούμε να επεκταθεί στα ιδιωτικά όχημα τουλάχιστον όχι τώρα. Τζιμ, μπορούμε να βάλουμε το κεφάλι σου στον Τουρβά, αλλά δεν θέλουμε να κάτσουμε εμείς. Ο κ. Ερτσοκ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ο κ. Ερτούκ, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Higgins για το έγγραφο εργασία, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι θέσει που υποστηρίζει. Και συμφωνώ απόλυτα με το γεγονό ότι τα κρατημέλη δεν εκτέλεσαν τα κατοίκοντά του, γιατί οι συνάδελφοι όντω. Γι' αυτό έχουμε τεράστια προβλήματα σήμερα, επειδή δεν ήταν τεθειμένα τα κράτη-μέλη στο παρελθόν να συνεργαστούν και δεν είμαστε πλέον τεχνικά στο σημείο που θα έπρεπε να είμαστε. Και αυτό πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συχνά. Να πω ότι πριν από το χειμερινό διάλειμμα είχαμε συμφωνήσει στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της διαλειτουργικότητας. Και αυτό λοιπόν συγκαταλέγεται στα θέματα διαλειτουργικότητας. Αν δεν συμφωνούμε και αν δεν το κάνουμε αυτό, προς τα που οδεύουμε να ρωτιέμαι. Άρα σας υποστηρίζω, συνάδελφε. Αυτό που θα ήθελα να θίξω είναι το κατά πόσο είτε αποφασίσουμε για διόδια είτε για αυτοκόλλητα, σίγουρα χρειάζεται διαλειτουργικότητα, είπαμε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να σκεφτούμε πού μπορούμε να δράσουμε ήδη σήμερα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα διόδια για τα φορτηγά. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα σε διάφορα ή σε όλα τα κράτη-μέλη να, να συμπεριλάβουμε, να εσωτερικοποιήσουμε το εξωτερικό κόστος στη δική μου χώρα, στη Γερμανία, η οποία α, πεισματικά αρνείται να εσωτερικοποιήσει στα για το εξωτερικό κόστος και αν ξέρουμε πόσο, πόσο ζημιά προκαλεί ένα φορτηγό και πόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η ζημιά που προκαλεί στο δρόμο το φορτηγό από ότι ένα ιδιωτικό όχημα, όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Κάτι άλλο που θα ήθελα να θέξω είναι Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε διάφορες μεταξύ... Ε, έχει απλευθεί η αγορά για τα ε, αστικά λεωφορεία, τα λεωφορεία μεγάλων διαδρομών και αυτό προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, δεν επιβάλλονται ε, τα ίδια στις δρομικές μεταφορές και στις μεταφορές με λεωφορεία. Επίσης, να μιλήσω για τα διόδια για τα γιοταχή, να σας ενημερώσω ότι η νομική υπηρεσία του Γερμανικού Κοινοβουλίου, του Γερμανικού Bundestag, γνωμοδότησε για το θέμα αυτό ακριβώς. όπου καταλήγει στο πόρισμα ότι δεν, ήταν, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διαφορετικέ επιβολέ διοδίων, διαφορετικά τέλη διοδίων για διαφορετικέ εθνικότητε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το είπε και ο κύριο Χίγκιν. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο θέμα αυτό. Το γεγονό ότι θα πρέπει να προσέξουμε και να λάβουμε υπόψη και τους ε, υπαλλήλου, ε, τους εργαζόμενους στις ε, περιφέρειες να σας πω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχουν τέτοιες διαφορές, γιατί ο κόσμος αυτός, ο οποίος δουλεύει σε περιφέρειες κοντά στα σύνορα, χρειάζεται το αυτοκίνητο. Και δεν θα καταλάβει, δεν θα κατανοήσει, γιατί θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβληθεί επιπλέον φόρος στο αγιοταχή. Ένα άλλο παράδειγμα στον τομέα αυτό, αν κατάλαβα σωστά, ή τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας, υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτού που χρησιμοποιούν ε, το δρόμο καθημερινά και από αυτούς που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο μία φορά την εβδομάδα. Και θα πρέπει να υπάρχει και διαφορά μεταξύ αυτού που οδηγεί την πόρσε και αυτού που χρησιμοποιεί ένα περιβαλλοντικά φιλικό αυτοκίνητο. Και σε αυτού, λοιπόν θα πρέπει να γίνει τη διάκριση στην επιβολή τελών διοδίων. Και επίσης να σας πω ότι η αρχή επιβολής διοδίων θα πρέπει να επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει διαλειτουργικότητα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί και πέρα μπορεί να, καταλα... να αποφασίσει κάθε κράτος μέλος τι θα κάνει. Μάικλ, θα μπορούσε να είσαι σύντομο γιατί φτάνουμε στο τέλος. Ναι, ο κύριος Κράμερ. Θα είμαι σύντομο. Εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστου. αποτελεί στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το πετύχουμε. Έχουμε ένα ανταγωνισμό μεταξύ λεωφορείων, ε, τρένων και οχημάτων, ιδιωτικών οχημάτων. Και ξέρουμε ότι αυτά που υπάρχουν σήμερα δεν επαρκούν. Έρωτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είχατε την πρόθεση να κάνετε πίσω στο σημείο αυτό σε ό,τι αφορά την επιβολή, το ύψος του επιβαλλόμενου διοδίου. Γιατί τελικά οδηγείται ο οδηγός σε μια απόφαση να πάρει ένα δρόμο που μπορεί να είναι πιο μακρύς, αλλά να έχει πιο χαμηλά διόδια. Εμείς κάναμε μια σχετική μελέτη με τους από τους πράσινους. σε ό,τι αφορά τα ποσά που επιβαβάλλονται στους ε, οδηγούς δυτικών οχημάτων στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Ήταν μια συγκριτική ανάλυση. Μιλάμε για τα ποσά που χρειαζόμαστε αλλά κανείς δεν κοιτάει αυτά πόσο αποτελικά επιβάλλονται στον οδηγό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραμίτσος, δεν ήξερα ότι έχετε ε, ηλεκτρονική υπηρεσία και λειτουργία, αλλά από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρώτον, να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν το λόγο σήμερα το πρωί, διότι πιστεύω ότι σωστές ήταν οι παρατηρήσεις λάβαμε υπόψη στις εκθέσεις. Μπορεί να βελτιώσουμε ωστόσο ακόμα το κείμενο και περιμένω την έκθεση του κ. Χίγγιντς γι' αυτό. Να πω καταρχάς ότι υπάρχει σήμερα η τεχνολογία, την έχουμε, που μας επιτρέπει πρώτον να επιβαρύνουμε βάση της θέσης του οχήματος, της απόστασης που, που διανύει, του χρόνου της ημέρας, της ε, εβδομάδας, του αν είναι καλοκαίρι ή όχι και της κατηγορίας του οχήματος που λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση, τον, το θόρυβο, τη ζημιά που προκαλεί. Υπάρχει λοιπόν τεχνολογία. Όταν ετοιμάσαμε τις προτάσεις μας το 2004 και μετά είχαμε και την απόφαση του 2009, πιστεύαμε ότι μέχρι τα 12 θα ήταν διαθέσιμες, ε, οι διαθέσιμες στοιχεία. Αυτή είναι η υποχρέωση και των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα. Δέκα χρόνια μετά, πέρσι δηλαδή, οι Αμερικανοί ήρθαν και είπαν μέχρι το 2015 το Κογκρέσο, το 2016, θα πρέπει να έχει υιοθετήσει ένα διαπολιτιακό σύστημα που θα λειτουργεί με τέλεια συνοχή. Γιατί δεν έγινε αυτά. Δύο λόγοι είναι Πρώτον, τα κράτη-μέλη δεν ήταν πρόθυμα να προχωρήσουν διότι είχαν περιοριστεί υπερβολικά από τους υπάρχοντες παρόχους των συστημάτων διοδίων. Και αυτοί πρέπει να, να τους μευθούμε διότι δεν θέλουν ε, να προχωρήσουν. Θέλουν την ε, εχμάλωτη αγορά τους και τίποτα άλλο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε δύο εναλλακτικέ λύσεις. Το μπαστούνι και το καρότο. Το μπαστούνι έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες παραπομπής 22 κρατών μελών γιατί δεν έχουν εφαρμόσει το σύστημα της διαλειτουργικότητας των διοδίων μέχρι τον Οκτώβριο πέρσι. Είπαμε ωστόσο ταυτόχρονα καλό είναι το μπαστούνι αλλά τι κάνουμε για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Και τι κάναμε. Ξεκινήσαμε με τακτικές συναντήσεις με τον ιδιωτικό τομέα και τα κρατημέλη για να ξεκινήσουν πιλωτικά συστήματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, τις βασικές, Ολλανδία, ίσως και Δανία, ξεκινώντας από ένα πυρήνα και επεκτηνόμενη με ένα σύστημα που θα είναι πλήρως διαλειτουργικό και θα επιτρέπει τη συνέχιση των διαδικασιών. Να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα διοδίων που θα υφίσταται. Υπάρχουν οι προδιαγραφέ και για χερσαίε και για δορυφορικέ επικοινωνίε. Δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει βούληση να προχωρήσουν προ ένα τέτοιο διαλειτουργικό σύστημα από πλευρά των άλλων. Γι' αυτό υπάρχει και ανακοίνωση. Περιμένουμε λοιπόν και από εσά να ξεκινήσετε τι πιέσει. Σα είπα ότι ξεκινήσαμε τι διαδικασίε, αλλά είναι σημαντικό, διαδικασία αλλά είναι σημαντικό και το Κοινοβούλιο να βοηθήσει διότι πρόκειται όντω για μια αποτυχία των εθνικών διοικήσεων και του ιδιωτικού τομέα να προχωρήσουν. Και αυτό που θέλουμε είναι να ξεκινήσουν τουλάχιστον περιφερειακά προγράμματα φέτο, όπω σα είπα είναι κομμάτι του καρότου. Είπαμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα ότι είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε ή να συγχρηματοδοτήσουμε το έργο αυτό για να διευκολύνουμε τι εξελίξει τη υπηρεσία σε όλη την Ευρώπη. Αυτό νομίζω είναι το πλαίσιο, το ιστορικό πλαίσιο. Θα επανέλθουμε στο ίδιο ζήτημα. Σημαντικό είναι ωστόσο να θυμόμαστε ότι στα ιδιωτικά οχήματα θέλουμε να εφαρμόζεται η αρχή της μη διάκρισης, δεν είναι σωστό. Είδαμε τις δυσκολίες ε, σε κάποια κράτη-μέλη που θέλουν να αντιμετωπίζουν τα εθνικά γιοταχή διαφορετικά από τα δαπά όταν το συζητούμε τα κράτη-μέλη, ε, το θέτουμε πάντα για να το αποφύγουμε. Επίσης είναι σημαντικό ε, ο αντιπρόεδρος Κάλλας μπορεί να προτείνει μια πρωτοβουλία για την επιβολή τελών στους δρόμους γενικότερα που στηρίζεται πάνω κάτω στην ε, αρχή της επιβολής τελών στη χρήση του δρόμου. Το είπατε ήδη κάποιοι από αυτό. Νομίζω ότι κράτησα το πεντάλεπτο, θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα, αλλά αν θέλετε καλύτερα είναι να επανέλθουμε για το μάτι όταν έχουμε την έκθεση του κυρίου Χίγκιντσα έτοιμη για παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μακαρμίτσο. Θε να προσθέσει κάτι Τζιμ? Όχι. Υπάρχει πρόταση, υπάρχει αποδοχή της πρότασης. Καλωσορίζω την υποστήριξη των σκιωδών, προσβλέπω σε μια στενή συνεργασία μαζί του. Επίση θα λάβουμε υπόψη τις απόψει των άλλων των μελών. Κάτι που θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι ότι δέχομαι τα σχόλια για την εμπιστευτικότητα. Το είπε ο κ. Μπένιον, το ευρύτερο θέμα τη πιθανή εκμετάλλευσης των δεδομένων. Εμεί θα εξασφαλίσουμε και μια βασική αρχή μα θα είναι να μην υπάρξει ακριβώ καμιά, καμία ε, κατάχρηση. Τώρα, για την ε, επιβολή διοδίων. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε στα κρατημέλη τι θα φορολογούν. Το κράτο μέλο θα αποφασίσει. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι η απλοποίηση. Το είπαν πολλά κρατημέλη. Η απλοποίηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προχωρούμε με την ε, πρόταση αυτή. Αν δείτε την κατάσταση τώρα, θα δείτε. Αν φύγει κάποιο από την Πορτογαλία και πάει στην Ολλανδία, έχει έξι διαφορετικά στοιχεία, εργαλεία, ε, μηχανάκια, βινιέτες που πρέπει να πληρώσει. Και η Επιτροπή το ίδιο λέει. Αν δεν το δούμε αυτό δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη ε, εμπορική εκμετάλλευση των ε, μηχανημάτων ή των δομών αυτών από τους χρήστε. Καταλαβαίνω τις επιφυλάξει του κ. Μπένιον, αλλά εγώ είμαι αποφασισμένος. Αυτό θα το πετύχουμε στην Επιτροπή τώρα και περιμένω τη βοήθειά σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Σας υποστηρίζει ο κύριος Μπένιον, αλλά θέλει να είσαι εσύ στην εμπροστοφυλακή, να μην είναι αυτό. Η έκθεση θα είναι έτοιμη στις 7 Μαρτίου, προθεσμία υποβολής των 20 Μαρτίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 23 Απριλίου. Μετά την εξέταση των τροπολογιών στις 22. Εντάξει. Προχωρούμε. Παρουσίαση της μελέτης για τα ΔΕΒ μείζωνα έργα από το Ινστιτούτο Φραγκοφ της Γερμανίας με τη συμμετοχή των εταιριών Kiden Prog από την Ελβετία. Ελάτε εδώ αν θέλετε. Okay, gentlemen. Okay, so. Λοιπόν, θα ξεκινήσετε εσείς ε, κύριε Σάντε φαντάζομαι. 15 λεπτά ο καθένας ομιλητής, ερωτήσεις και απαντήσεις για να τελειώσουμε στις 12.30. Ο κύριος Σάντε από το Φράνχοφ Institute Ξεκινήστε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλημέρα. Θα σας μιλήσω για το έργο μας TEN ΔΕΛΤΑ ε, επενδύσεις και δαπάνες. Είναι γνωστό για σας. Αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων Ξεκινήσαμε στη δεκαετία του 90. Τα προγράμματα έργα αυτά είναι μεγάλα έργα. Είχαμε πολλές φάσεις ανάπτυξής τους που συνδέονται και με διάφορες, διάφορα στάδια οδηγιών για την υλοποίησή τους. Είχαμε τις οδηγίες του 96 πρώτα, κατόπιν του 2004 μια ενημέρωση και μια αναθεώρηση το 11 που συζητείται αυτή τη στιγμή εδώ για το οποία γίνεται η μελέτη. Το αντικείμενό της ήταν να συζητήσει και να εντοπίσει επιχειρησιακά προβλήματα που συνδέονται με την αξιολόγηση των μεγάλων έργων, να παράσχει συστάσεις για το πώς ε, αυτά τα προβλήματα που συνδέονται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα μπορούσαν να μετριαστούν ή να επιληθούν. την ομιλία μας την ε, χωρίσαμε σε δύο τμήματα. Πρώτον, μελέτες περιπτώσεων. Είχαμε κάνει δέκα μελέτες περιπτώσεων. Θα σας μιλήσω για τα ευρήματα και κατόπιν θα μπούμε στο δεύτερο τμήμα. Πώς είναι η κατάσταση της μοντελοποίησης και της αξιολόγησης έργων. Αυτό είναι το αντικείμενο μου. Η μελέτη έγινε πρώτον με ανάλυση της βιβλιογραφίας για την αξιολόγηση τέτοιων έργων, ιδίω μεγάλων έργων. Κατόπιν εντοπίσαμε και ορίσαμε κριτήρια επιλογής για τις μελέτες περιπτώσεων μαζί με το προσωπικό του Κοινοβουλίου και επιλέξαμε 10 μελέτες περιπτώσεων για την έρευνά μας. Η ανάλυση περιλάμβανε και επιτραπέζια έρευνα, δηλαδή κόστος, όφελος, προβλέψεις, αλλά και επιτόπια έρευνα, συνεντεύξεις με τους εμπλεκόμενους φορείς ε, από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους υπεύθυνους των διαφόρων έργων. Αυτό κάναμε. Βάσει αυτών των δύο βρήκαμε Συστάσει και αναπτύξαμε, ε, βρήκαμε συμπεράσματα και αναπτύξαμε συστάσει. Οι δέκα μελέτες περιπτώσεων που εν τέλει επιλέξαμε περιλαμβάνουν 5 σιδεοδομικά έργα. Μην ξεχνάτε ότι μεγάλο, μεγάλος αριθμός των έργων ε, που εξετάζουμε είναι σιδεοδομικά που είναι πιο μεγάλα έργα. Υπάρχει ένα μεικτό οδικό σιδεδομικό, δύο οδικά ένα ε, ποτάμιον μεταφορών. Επίσης είχαμε το καθήκον να εξετάσουμε περιπτώσεις εξπόστο, να συμπεριλάβουμε δηλαδή περιπτώσεις εξπόστο όπου θα ήταν δυνατό να εξετάσουμε και τον προγραμματισμό αλλά και εξπόστο βρήματα, πώς δηλαδή ο προγραμματισμός ε, υλοποιήθηκε εν τέλει, ποια ήταν η έκβαση όπου κάναμε έξι εξπόστ μελέτες περιπτώσεων και τέσσερις ε, μελέτες περιπτώσεων που βρίσκονται σε φάση προγραμματισμού αυτή τη στιγμή και που αποτελούν μέγα έργα, με τεράστια έργα, κομμάτια αυτών των ε, διευρωπαϊκών δικτύων. Θα δείτε στη διαφάνεια αυτή επίσης ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε μια περιφερειακή ισορροπία. Έχουμε έργα και στην Ευρώπη των 15, αλλά και έργα που προγραμματίζονται ή, εφαρμοζούνται και στις νέες 12 χώρες της Ένωσης. Τώρα, για τα ευρήματα. Για το κόστος των έργων και την αξιολόγησή τους. Δέκα μελέτες είχαμε με κόστος 100, από 131 εκατομμύρια ευρώ έως 2,4 δις. Η μικρότερη μελέτη αφορούσε ένα οδικό πρόγραμμα τον ε, Α11 Βερολίνο-Πολωνία και το μεγαλύτερο έργο είναι η μελέτη για την, ε, το συνδεδομικό δίκτυο της δυτικής ακτής 2,4 δις. Αυτή η γραμμή περιείχε δύο μελέτες περιπτώσεων. Η πρώτη αφορούσε την, ε, μια πρώτη φάση που οδήγησε σε απόφαση του 1994 όπου βρήκαμε το αρχικό κόστος του έργου, δύο δις περίπου, και που περιλαμβάνει η υλοποίηση 2,4 δις. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε το 2003 με αναθεώρηση του σχεδίου και νέο προγραμματισμό που είχε κόστος, προσδοκόμενο κόστος 11,8 δις και που έφτασε στα 12,4 τελικά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είχαμε μεγάλη αύξηση. Στην τρίτη στήλη, στην τέταρτη στήλη μάλλον, στην τρίτη στήλη το BCI είναι Benefit Cost Restraints. Εδώ εντοπίζουμε ε, συντελεστές κέρδους κόστους. Είδαμε ότι εκεί υπήρχαν από χαμηλό μέχρι 6,5 Μία παρατήρηση πρέπει να κάνουμε για αυτό το συντελεστή κέρδους κόστους. Ε, ο συντελεστής εξαρτάται πολύ από την επιλεγόμενη περίοδο αποπληρωμής. Το 1,9 που έχουμε στο, στο Brenner επιτεύχθηκε με η κοινωνική έκπτωση 55%. Ε, η αξία είναι καθαρή τρέχουσα αξία. Μόνο για την βασική γραμμή της Δυτικής Αρχής υπάρχει εκτίμηση για 190 εκατομμύρια στερλίνες καθαρή παρούσα αξία και η οικονομική αξιολόγηση στηριζόταν και στην περίοδο βέβαια αποπληρωμή, όπως σας είπα. Εντοπίσαμε δηλαδή έργα που είχαν εκτιμόμενη περίοδο πληρωμής από 7 έως 20 έτη. Για το άλλο, τα άλλα σημαντικά στοιχεία των νέων καθοδηγητήριων γραμμών που συζητήθηκαν και στο Κοινοβούλιο, τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, το EIA, η προτελευταία στήλη, είδαμε ότι σχεδόν όλα, σχεδόν όλες οι προσεγγίσεις είχαν κάποια μορφή περιβαλλοντικού αντικτύπου, διαφοροποιημένη βέβαια ανάλογα με το, ως προς το περιεχόμενο και εξαρτώνταν από την περίοδο υλοποίηση. Η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου που γινόταν στη δεκαετία του 90 δεν πληρούσε τα κριτήρια που απαιτούνται ε, τώρα. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η, κλιματική, η, η μελέτη αντικτύπου για το κλίμα. Υπήρχαν στη, στις μελέτες στο παρελθόν θεωρητικά, αλλά στην πράξη πολλές πολλά από τα έργα δεν είχαν τίποτα. Προσοχή βέβαια, δεν υπάρχει ορισμός του τι ονοούμε μελέτη κλιματολογικού αντικτύπου. Δύο έργα είχαν μία αξιολόγηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της κίνησης. Αυτό είναι ένα τμήμα της μελέτης κλιματολογικού αντικτύπου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνονταν τέτοιες μελέτες και σε άλλες ε, απλές μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου. Τώρα, οι μελέτες ε, περιπτώσεων που κάναμε ανάλυση ex post. Έξι ήταν, όπως σας είπα. Περιμέναμε ήταν έξι, ναι. Πρώτον, πρέπει να, να διακρίνουμε μεταξύ τριών διαφορετικών τύπων κόστους. Υπάρχει καταρχάς το αρχικό κόστος, όπως το αποκαλούμε. Το κόστος που προϋπολογίστηκε στο ξεκίνημα όταν ξεκίνησε ο προγραμματισμός. Για τη γραμμή Μπετούβε ήταν 1,5 δις. Αυτή, αυτό το κόστος, όταν προτάθηκε η ιδέα. Κατόπιν ξεκίνησε ο προγραμματισμός Εξετάστηκαν άλλες διαστάσεις ε, του κόστους, Φερρυπίν η δημιουργία σειράγκων, ε, το περιβαλλοντικό αντίκτυπος γενικότερα. Οπότε αυξήθηκε στα 3,6 δις. Και αυτή ήταν η απόφαση αυτό ήταν ο υπολογισμό πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η απόφαση να χτιστεί η γραμμή Μπετούβε. Υλοποιήθηκε το 2007 και το κόστος, το τελικό κόστος ήταν 4,7 δις. Για να το συγκρίνετε τώρα, το κόστος είναι ε, ξεπέρασε τον προπολογισμό κατά 27% αυτό το overrun που λένε παίρνεις ε, το πραγματικό κόστος από το αρχικό κόστος και βλέπεις ότι υπάρχει μια πόσο σημαντική είναι η υπέρβαση κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε για τη διαφάνεια αυτή βρήκαμε ότι σε δύο μελέτες περιπτώσεων δεν είχε γίνει ολοκλήρωση. Η... Το 7 και το 8, ο, ο δρόμος σεβιλιου Έλβα και το δρόμος Βερολίνο Πολωνία. Εμεί είχαμε ξεκινήσει επιλέγοντα αυτά διότι είχαμε τα στοιχεία τη Επιτροπή, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα παρακολούθηση τη ε, πρόοδου στα έργα αυτά είδαμε τις επίσημες δηλώσεις, αλλά όταν δίδαμε μετά τις λεπτομέρειες διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση ήταν διαφορετική από τα επίσημα κείμενα. Κατόπιν προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ένα σχέδιο, ένα σχήμα για την διαδικασία απόφασης για, τα, για τη συγχρηματοδότηση. Αυτή είναι η ιδανική διαδικασία, αλλά βοηθά να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα κατά τη διάρκεια λήψη απόφασης. και να αντιμετωπίσουμε όλες τις πιθανές αιτίε υπέρβασης κόστους. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω βέβαια όλο τον πίνακα εδώ, γιατί θα σας φάω μια ώρα. Απλά να τονίσω κάποια θέματα υπάρχουν τρία κουτάκια που δείχνουν τα σημαντικά σημεία της απόφασης. Δεν, μπορώ να, δεν μπορείτε να τα δείτε. Πρώτον, το έργο πρέπει να προταθεί. Για τη γραμμή Μπετούβε, για παράδειγμα, υπήρχε το αρχικό πλάνο που ήταν η πρόταση του έργου και κατόπιν έγιναν οι πρώτες μελέτες που τις λέμε μελέτες προ σκοπιμότητας. Να σας πω για παράδειγμα, ε, τούνελ, γέφυρα, τούνελ και γέφυρα, αυτή είναι η δεύτερη φάση του προγραμματισμού. Κάνουμε δηλαδή μία μελέτη αντικτύπου με τις διάφορες εναλλακτικέ και φτάνουμε σε συμπεράσματα για το ποια από τις δύο είναι η προτιμητέα. μετά το βάζει στη μελέτη, στη μελέτη υλοποίησης και εξετάζεις τις διάφορες αναλλακτικές οδούς. Πάλι εδώ μπορείς να κάνεις ε, λεπτομεριακές μελέτες, ξέρεις ποιες είναι οι εναλλακτικές οδοί και μπορείς να λάβεις την τελική απόφαση γνωρίζοντας τις Εναλλακτικέ δυνατότητες. Αυτό είναι κάτω δεξιά. Και με βάση την απόφαση για το έργο παίρνει την απόφαση για τη χρηματοδότηση. Αυτό το, το σχέδιο, αυτή, αυτή η απεικόνηση θα οδηγούσε κανονικά σε μια καλή επιλογή του έργου. Ένα στοιχείο που είναι κρίσιμο στη διαφάνεια αυτά είναι ο προγραμματισμός ε, μεταφοράς κάτω αριστερά. Ε, η πρόβλεψη δηλαδή μεταφορικού όγκου, κάτι που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη και είναι καθοριστικό για τη βιωσιμότητα του έργου. Ε, μερικές φορές υπολογίζουν, υπε, υπερβάλλουν ως προς την πρόβλεψη μεταφορικού όγκου και δεν μπορούν ποτέ να αποπληρώσουν. Τα συμπεράσματα των μελετών περιπτώσεων. Κάποια να τονίσω. Πρώτον, τι εντοπίζουμε. Πρώτον, η έλλειψη σαφούς ορισμού, σαφούς καθαρού ορισμού του έργου δημιουργεί υπερβάσεις. Αυτό το είδαμε και στο παρελθόν και σε μελέτες που συνεχίζουν τώρα, Φερρυπίν, το Rail Baltica, που δεν έχει ακόμα σαφή καθορισμό. Ήδη αναφέραμε την ε, πρόβλεψη μεταφορικού όγκου, πιθανή πηγή αποτυχιών ε, στην χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός έργου. Ένα πρόβλημα που δεν ανέφερα είναι ανάγκη διαφάνειας για το έργο, τόσο ώστε οι μελέτες ε, που περιγράψαμε να γίνονται δημοσία, με συζήτηση και συμμετοχή του κοινού. Η κατανόηση του έργου μειώνει τους κινδύνους να υπάρξουν προβλήματα μετά τον προγραμματισμό και όταν έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή. Κάτι άλλο. Η ενημέρωση για τα διάφορα έργα είναι κατακαιρματισμένη. Πρέπει, κάποια τα βρίσκει στην Επιτροπή, μιλάς με Υπουργεία. Είναι πραγματικά δύσκολο να έχεις όλα τα δεδομένα στοιχεία. Αυτά. Και τώρα θα το δώσω στον συνάδελφο. Θα το λόγο στον συνάδελφο. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι. Με αυτό το τεχνολογικό και καταρχάς θελήσαμε να μελετήσουμε τις μεθόδους αξιολόγησης που εφαρμόζονται για τα μείζωνα έργα υποδομή στον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζοντα, θα κάνω γενικέ παρατηρήσει και θα συνοψίσω. Τι ακριβώ κάναμε. Πρώτα απ' όλα, η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έργα μπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις. Στο φάση σχεδιασμού και στη φάση εφαρμογής, όταν πρόκειται για συγχρηματοδότηση και θα πρέπει να καταβληθεί ένα μέρος του δαπάνη κράτη-μέρη. Τώρα, σε σχέση με την τη συνδυναξία αυτών των δύο φάσεων. Πρέπει να πούμε ότι στη φάση σχεδιασμού υπάρχουν ε, κάποια θέματα που επηρεάζουν τα κράτη-μέλη στις αποφάσεις τους, ότι πιστεύουν ότι θα συγχρηματοδοτηθούν. Πράγμα το οποίο επηρεάζει το όλο σχέδιο. Και πολλές φορές στην φάση του σχεδιασμού μπορούν να υπάρξουν αποτυχίες. Στην πρώτη φάση έχουμε τρία επίπεδα. Στρατηγική για την ε, θέση των στόχων και την παγιωσή τους. Δεύτερον, ανάπτυξη του σχεδιασμού του δικτύου, δηλαδή πολυκομβικό δίκτυο το οποίο θα είναι το κατάλληλο για να μπορέσουν ε, να υλοποιηθούν οι στόχοι. Τρίτο επίπεδο, το επίπεδο του project, του σχεδίου που θα επιλεγεί και σχεδιασμός του. Και στη, πρέπει να πω ότι εν μέρη αλλάζει όλη η διαδικασία με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι γίνεται προσπάθεια να συνδυαστούν διάφορα σχέδια, projects, πράγμα το οποίο έγινε όταν έγινε η εφαρμογή των πρώτων δικτύων ΔΕΔ, το 2004 ήδη. Τρίτο επίπεδο. Πέρασε πριν από το πρώτο της στρατηγικής που ήρθε στην τρίτη σειρά και έπρεπε να μελετηθεί αν υπήρχε προσθέμενη αξία σε αυτό το πρόσχερο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές επιτυχίες. Κακό σχεδιασμός, καλκοί ορισμοί. Και πολλές φορές ε, έγινε αλλαγή των προτεραιότητων των στόχων και των επιπέδων. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή αλλάζει και όλα αυτά έγιναν στα πλαίσια της Λευκής του 2011. Πρώτα λοιπόν πρέπει να γίνει ο ορισμός του σχεδίου και σήμερα η βάση ε, για την ανάπτυξη των ΔΕΔ είναι οι κατάλληλοι και έτσι αποφεύγονται πολλά από τα λάθη τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει δεν θα πω σε λεπτομέρειες όσον αφορά αυτά τα ασφάλματα. Θα σας αναφέρω όμως κάποιες συστάσεις. Δεν θα αναφέρω την μεθοδολογία. Είναι κρίμα γιατί εγώ είμαι ερευνητή. Και με μεγάλη ευχαρίστηση θα έκανα και όσον αφορά την μεθοδολογία κάποιες ε, κρίσεις και παρατηρήσεις για τις αποτυχίες, για τις λάθος επιλογές, αλλά πάση περιπτώσει θα κάνω κάποια θα φτάσω σε κάποια γενικά συμπεράσματα, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αρχίσουμε με ένα σχέδιο τη στρατηγικής και με ένα σαφές, ε, σαφή ορισμό του σχεδίου το οποίο ε, θέλουμε να αναπτύξουμε. Δηλαδή, master plan κατάλληλο. Δεύτερον, να συνεχίσουμε με την ε, μεθοδολογική ανάπτυξη του προτύπου μεταφορών που θέλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή. Και παίρνω το κατάλληλο ε, παράδειγμα για τον αυτοκινητόδρομο στη Σεβίλη. Εκεί είδαμε ότι δεν είχε γίνει η κατάλληλη ανάπτυξη του σχεδίου. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικό της σύστημα ελέγχου αλλά τα κράτη-μέλη χρειάζονται για ένα ευρωπαϊκής κλίμακας έργο κάποιες συγκριτικές μελέτες και αναλύσεις για να μπορέσουν να καταλάβουν τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάποια μικρή χώρα δεν θα πρέπει να υφίσταται κυρώσεις για μεγάλα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν για μια άλλη χώρα. Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν και με τις προσδοκίες και τις ε, εκτιμήσεις κάθε χώρας. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη μελέτη ε, κόστους απόδοσης και να λαμβάνεται υπόψη και οικονομικές εξελίξεις. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Τρίτη παρατήρηση. Να δοθεί βοήθεια ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα διάφορα κριτήρια τα οποία θα ακολουθηθούν, κυρίως στις νέες χώρες μέλη. Αυτό είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν διάφορες συμβουλευτικές ομάδες, οι Jaspers, για να βοηθήσουν αυτές τις ναι, χώρες να κατανοήσουν περί τίνος πρόκειται. Και εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την στρατηγική ε, που θα ακολουθηθεί, τις ε, μελέτες επιπτώσεων για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά μπορούν να συμπεριλάβουν και το σύνολο όλων των ενιών στα πλαίσια του AA, του CA και μόνο για θέματα εκπομπής αερίων είναι η επιπτώση με τον πιο ενοποιημένος. Επίσης, θα πρέπει να αναπτύξουμε μία πιο ε, λεπτομεριακή προσέγγιση για να αξιολογήσουμε τις δευτερεύουσες επιπτώσεις και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για, τις, ε, για τα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα τις αξιολογήσεις, τις εκτιμήσεις, τις ε, κάνει η Κομισιό. Αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι και σε Ευρωπα... σε επίπεδο κρατημένου. Μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί ο ορισμός, ο σαφής ορισμός και δεν έχει μετρηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είναι κάτι το οποίο ε, αναφέρεται, αλλά δεν έχουμε ένα πρότυπο, ένα μοντέλο για να μπορούμε να έχουμε μια πιο ε, πρακτική ε, και πραγματιστική έννοια. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα σχέδια να λαμβάνουν υπόψη αυτά τα στοιχεία, να λαμβάνουν υπόψη επίσης τις, ε, ε, τα οικονομικά προβλήματα, την οικονομική κρίση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο ε, σχεδιασμού, αλλά και να ληφθεί υπόψη όταν, όταν μιλούμε για συγχρηματοδότηση. Και τέσσερις συστάσεις τώρα που έχουν σχέση με τη φάση εφαρμογής είναι πρωταρχική σημασία να δούμε κατά πόσον τα, να, είμαστε σίγουροι ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται θα είναι ποιοτικά. Η διαφάνεια και οι κοινοί όροι που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται θα πρέπει να καθοριστούν. Θα πρέπει να εναρμονιστούν οι κανονισμοί χρηματοδότησης. Να ξέρουμε οι χρηματοδότηση και το ύψος των κονδυλίων να καθοριστούν. Ο συντονισμός και η διαφάνεια είναι πρωταρχική σημασίας και θα πρέπει να υπάρχει ένα, ε, να συσταθεί ένα κεντρικό γραφείο συλλογής δεδομένων για τα σχέδια τα οποία θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Μπορούμε όλα αυτά τα δεδομένα να τα πάρουμε από τους υπεύθυνους τον ΔΕΔ σε κάθε χώρα, αλλά η διαφάνεια, κατά την άποψή μας, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού στο μέλλον. Και τελικά, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, για τα μείζωνα έργα είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων σε όλα τα στάδια. Ακόμη και ευθύ εξ αρχή να υπάρχει συμμετοχή ενώσεων πολιτών ώστε να ξέρουν περί τίνος πρόκειται για να μην καταλήγουμε όταν βρισκόμαστε στη φάση ανάπτυξης σε προβλήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν και στη δικαιοσύνη και στα δικαστήρια όπως είδαμε σε ένα από τα προβλήματα στις περιπτώσεις με τη Γερμανία. Θα πρέπει λοιπόν από την πρώτη φάση του προγραμματισμού μέχρι της εκτέλεσης να είναι ε, εξασφαλισμένη συμμετοχή όλων των ε, ενδιαφερομένων φορέων. Συνάδελφοι τώρα έχουν το λόγο. Κύριος Κάντσι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Είναι σημαντικό η Επίτροπή μας να ενημερώνεται για τέτοιου είδους ε, θέματα και θέλουμε και εμείς ότι κάνουμε να είναι ορατό σε όλους. Μιλήσατε για την ε, διάρκεια όλων αυτών των σχεδίων. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για θέματα προσθεμιών και εξουσιοδότησης για τέτοιου είδους έργα. Πρόκειται για σημαντικά θέματα, αλλά αν δεν υπάρχει και ασφάλεια για τους, τους επενδυτές, δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο. Αυτό είναι ένα πρωταρχικό σημείο κίνησης, εάν ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τέτοιου είδους εταιρικέ σχέσεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα ε, γίνουν πραγματικότητα, δεδομένου ότι ξέρουμε πόσο λίγα κονδύλια πλέον διαθέτουν οι κρατικοί προϋπολογισμοί. Τώρα, η οικονομική και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι εξίσου σημαντική για τέτοιου είδους έργα. Και κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ της αρχής και του, από την αρχή ως το τέλος. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή την ε, συνεκτικότητα, διότι τέτοιου έργα δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως μη συνεκτικά και ίσονος ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε από την αρχή ότι πρόκειται για σημαντικά έργα. Και εκτός από την υλοποίησή τους, θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε παρόντες σε όλες τις φάσεις για ενθάρρυνση, για προώθηση ε, της ποιότητας των έργων αυτών. Και για το όφελός τους γενικότερα για την κοινωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε, να προσελκύσουμε και άλλα κονδύλια από διαφορετικές πηγές για να κινητοποιήσουμε τα απαραίτητα κεφάλαια. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια. Ότι δεδομένου ότι έτσι έχουν τα πρότυπα τα οποία ακολουθούμε για να υλοποιήσουμε τα σχέδια αυτά και τα έργα αυτά τα μείζωνα, θα πρέπει να έχουμε μία λογική που θα μας επιτρέπει να ζητήσουμε και να επιτύχουμε την συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή μάλιστα, του ιδιωτικού τομέα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα αντέξουν στο χρόνο αυτά τα σχέδια. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά πρέπει να ανταποκριθούμε. Ευχαριστώ. Ο κ. Σέρτου, ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σάντα και τον κύριο Πενκάταρ για τις ε, πολύ χρήσιμες ε, πληροφορίες που μας έδωσαν. Είναι γνωστό νομίζω ότι το θέμα των ε, μεγάλων αυτών project είναι πολύ σημαντικό και προκαλεί έντονα συναισθήματα και στη Γερμανία. Θεωρούμε ότι ίσως να υπάρχει ένας ε, κορεσμός ο οποίος να ε, οδηγεί σε διαφορετική αντιμετώπιση από τις άλλες χώρες που υπάρχει ανάγκη ανάπτυξη υποδομής ε, συνεπάγεται τεράστιο κόστος και είναι και τεράστια και η πολιτική ευθύνη λοιπόν. Γιατί η πολιτική αυτή είναι αυτή που καθορίζει που θα χτιστεί τι. Με τον συνάδελφο Κουμουτσάκο θέλουμε να θέσουμε κατευθύνες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και έχουμε αναφέρει τα στοιχεία αυτά. Να αναφέρω και κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία. Καταρχάς, σημαντικό είναι να τεθούν στρατηγικοί στόχοι. Με πιο σαφή τρόπο. Κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλο έλλειμμα σήμερα σε ό,τι αφορά το συντονισμό των εθνικών ε, σχεδίων. Υπάρχουν κατάλογοι με τα project, αλλά χωρίς συντονισμό. Και η πληροφορία επίσης, οι πληροφορίες, η ενημέρωση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα δεν είναι συντονισμένη. Και αυτό θα πρέπει να τα προσέξουμε. Χρειαζόμαστε επίσης σαφή κριτήρια στην επιλογή και εφαρμογή των διαφόρων αυτών έργων. Επίσης, ανάλυση κόστους και ωφέλειας. Και αυτά θα πρέπει να εναρμονιστούν. Στις 18 Δεκεμβρίου το ψηφίσαμε μεγάλη πλειοψηφία. Ανάλυση κοινωνική κόστους και όφελους. Με μελέτη αντικτύπου και για το περιβάλλον και για το κλίμα. Αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να δικαιολογούμε τέτοια μεγάλα έργα. Χαίρομαι που, θέσατε θέματα και έλλειψης διαφάνειας σε ό,τι αφορά τα project αυτά, σε ό,τι αφορά τα έργα αυτά και στη φάση σχεδιασμού και στη φάση εφαρμογής αλλά και στο κόστος και στη λήψη απόφασης δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Υπάρχει το TNT Agency, η αρχή αυτή. Ίσως εκεί θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν μια συνολική εικόνα. Τελευταίο σημείο, το πιο σημαντικό για μένα, στην έκθεσή μας. Έγκαιρη και δεσμευτική συμμετοχή περιφερειακής και τοπικής ε, κοινωνίας και τοπικού επίπεδου. Αυτό δεν έχει συμβεί. Και ιδιαίτερα σε χώρες διαμετακόμισης υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίσης, αναφέρθηκαν τα εργαλεία trans. Trans tools. Σημαντικό εργαλείο, το οποίο δεν είναι γνωστό ιδιαίτερα. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί όμως. Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μήπως θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν σήμερα για ποιο λόγο δεν έχει συμβεί αυτό, πώς μπορεί να βελτιωθεί και ποια είναι η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορούν κάπου να συλλεχθούν τα στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη για μελλοντικά έργα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις που δώσατε. Συμμερίζομαι απόλυτα ένα μέρος της μελέτης, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος ένας από τους συζητές για τους νέους προσανατολισμούς των ΔΕΔ παρουσιάσαμε από την ομάδα κάποιες παρατηρήσεις ώστε να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον ορισμό, την εκτέλεση και τον εντοπισμό των κριτηρίων που χρησιμοποιούν τα διάφορα κράτη-μέλη για να καθοριστούν τα σχέδια τα οποία θα πρέπει να έχουν μια καθαρά ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Από όλες τις εξηγήσεις που δώσατε, Συμφωνώ ότι όντω θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και από αυτού να σα πω ότι η ομάδα μου κατέθεσε μία από τις τροπολογίες που ζητούσε και απαιτούσε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια όλων των αιτημάτων των κρατών μελών για όλα τα σχέδια και πλήρης διαφάνεια για τα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, επιθυμεί να χρηματοδοτήσει κάποια από τα σχέδια αυτά. Εγώ είμαι από αυτές που είχε ένα τρομερό πρόβλημα το οποίο δεν μπόρεσα να επιλύσω. Δηλαδή ήθελα να ξέρω για ένα θέμα προτεραιότητα που με ενδιαφέρει, ποιε είναι οι αποφάσει που ελήφθησαν σε πρώτη φάση, ποια ήταν τα κριτήρια επιλογή ή απόρριψη, ποια ήταν η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κράτους μέλους. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας πλήρης διαφάνεια. Και θα ήθελα επί του θέματος να σας ερωτήσω το εξή. Στη διάρκεια όλες αυτές τις διαδικασίες και των αναλύσεων που κάνετε, δεν αναφέρατε τουλάχιστον ε, ορίσατε, αξιολογήσατε μάλλον το ρόλο των ε, Ευρωπαίων συντονιστών για να μπορέσετε να κάνετε σαφείς τους ορισμούς βάσει των οποίων ε, προχωρείτε. Επίσης, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πώς αξιολογείτε τη συμμετοχή των περιφερειών στις χώρες τις οποίες έχουν αρμοδιότητες εκτελεστικές οι περιοχές και τα τοπικά όργανα. Κάτι το οποίο επίσης δεν κατάλαβα ίσως καλά τι γίνεται με το σχέδιο Βερολίνου-Πολωνίας και Σεβίλης-Ουέλβα. Είπατε ότι είχατε ε, διαφορετικές πληροφορίες. Τι συμβαίνει ακριβώς. Και βεβαίως συμμερίζουμε απόλυτα την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, καλύτερος συντονισμός και συμμετοχή των πολιτών. Από τις αναλύσεις που κάνετε όλων αυτών των σχεδίων μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα, παράδειγμα βέλτιστης ευρωπαϊκής πρακτικής. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τους εισηγητές για τις πληροφορίες που μας έδωσαν και τη μελέτη που έκαναν. Ήθελα να είδα τα κριτήρια επιλογής που κάνετε στην αρχή και ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα μόνο. Στην επιλογή αυτή υπήρξε, όπως είπε και η κυρία Μπιλμπάου, ένας εντοπισμός καλών και κακών πρακτικών. Έργα για τα οποία εμφανίστηκαν προβλήματα, για τα οποία δεν εμφανίστηκαν, πέραν των κριτηρίων που αναφέρθηκαν εδώ ή όχι. Επίσης, αναφέρεται ότι είναι μεγάλα έργα που έχουν προϋπολογισμό επταετίας, πολυετή, που δεν καλύπτει καν ε, μερικές φορές τις ε, προσδοκίες ε, δουλειά. γιατί στα έργα λένε α πούμε ότι θα κρατήσει τόσο. Ξεκινάμε από ένα προϋπολογισμό εμείς έχουμε έναν προϋπολογισμό που θα γίνει από το 2014 2020 ενώ έχουμε άλλους προϋπολογισμούς που φτάνουν ε, στα έργα αυτά το 2030 και το 2050. Λάβατε υπόψη αυτή την απόκληση. Είπατε επίσης ότι κάποιες χώρες ε, είναι πιο αισιόδοξε, κάποιε πιο απεσιόδοξε ό,τι αφορά τι οικονομικέ προοπτικέ. Εγώ ρωτώ, εσεί ω εμπειρογνώμονε μπορείτε να εντοπίσετε να κάνετε προβλέψεις για την υφιστάμενη κρίση. Λέτε ότι δεν υπάρχουν εργαλεία προσαρμογής σε περίπτωση μεγάλης κρίσης. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Τέλον, τέλος, διασυνοριακά έργα. Τι δυσκολίες βρήκατε. Ποιες είναι οι διαφορές νομοθετικού χαρακτήρα, Φερρυπίν, για, την, για τους διαγωνισμούς, για την υλοποίηση, για το επίπεδο ασφάλεια, για την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριος Κράμερ. Και εγώ ευχαριστώ φυσικά τους ομιλητές για την παρουσίαση. Μερικές ερωτήσεις για την επιλογή των έργων. Προφανώς και χρειάζεται γιατί όμως ε, το Eurotunnel που ήταν καταστροφή δεν επιλέχθηκε. Πώς ε, αποφασίζονται αυτά για το Femabelt. Το τούνελ προς τη Δανία μπορεί να μην παίζει κανένα ρόλο στη Γερμανία από την άλλη πλευρά. Αυτό λαμβάνεται υπόψη είναι αυτό, για παράδειγμα για το Τωρίνο. 12 εκατομμύρια, 12 δισεκατομμύρια. Κάποιοι εκτιμήσαν 28 εκατομμύρια, 36 εκατομμύρια. Συναντήθηκε ο Μάουρο Μόντι και ο Λαντ και αποφάσισαν να γίνει μέχρι συγχρηματοδότηση. και μόνο αυτό να συγχρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 40% μπορεί να ξεχάσει τα υπόλοιπα έργα. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στην εφημερίδα αναφέρεται ένα άρθρο για τη Φραγκφούρτη σε ό,τι αφορά τέτοιες συμπράξεις, αλλά και σε άλλες χώρες. Αναφέρεται ότι είναι κρυφές πιστώσεις για να αποφευθεί ε, η φραγμή χρέωσης. Οι συγκληματοδοτήσεις αυτές είναι ασφαλώς ε, κάτι το οποίο τελικά παίρνει πολύ πιο πολύ χρόνο και πολλά πιο πολλά χρήματα. Και σημαντική είναι και η σύγκριση. Για παράδειγμα έχουμε το διάδρομο της Βαλτικής και της Αδριατικής. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε διαλέξει άλλες οδούς που θα ήταν πιο οικονομικές. Ξέρουμε ότι ακόμα και στις μελέτες χρησιμοποιούνται πολλά κόλπα. Αυτά που θέλει η πολιτική τα δικαιολογεί με όποιο τρόπο βρίσκει. Αυτά που δεν θέλει θεωρεί ότι είναι πολύ ακριβά. Τελευταίο στοιχείο. Στο Βαρολίνο, στη Γερμανία, μεταξύ Νινεμβέργη και Ερφούρτης, έναν διάδρομο με 12% συγχρηματοδότηση. Αλλά δεν έχει κανένα ευρωπαϊκό αντίκτυπο αυτός ο διάδρομος. Πείτε μας, είναι 30-20%, 2-3%. Η συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. συνάδελφοι. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα κάθε φορά σε τέτοιες μελέτες, αλλά δεν δίνουμε αρκετό χρόνο στους ομιλητές μας για να μου απαντήσουν. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε το λόγο, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομος για να ζητήσω μετά από τους διδάκτορες να μας απαντήσουν στις απίστευτα πολλά ερωτήσει που ακούσαμε. Ο κ. Ρόιτερς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Δείτε την τελευταία παράγραφο των συμπερασμάτων πρώτα πρώτα. Η απόφαση, η διαδικασία λήψη αποφάσεων για τα δικτύα βελτιώθηκε σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω με τον καθορισμό των βασικών ε, ενιών και των διαγωνισμών ε, για την καθώς και τις τροποποιήσεις που θα υποβάλει σχετικά το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ. Η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει τους, μελέτε, τους ε, συντάκτες της μελέτης για το σύντομο διάστημα που το έκανε και τη γραμματεία της Επιτροπής που ετοίμασε τη μελέτη αυτή δύσκολη και διαφορετική από αυτή που είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια. Κάποιες παρατηρήσεις και να δώσω και μία απάντηση για τις παρατηρήσεις. Ένα από τα συμπεράσματα που αναφέρεται στη μελέτη είναι ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αρεσιμότητας και ε, αναλογικότητας. Αν ε, θέσουμε, αν χρηματοδοτούμε κατά 10% προφανώς δεν μπορούμε να θέσουμε πολύ λίγες προϋποθέσεις. Είδατε ωστόσο ότι εν γέννη αυξάνονται οι προϋποθέσεις. Επίσης, δεν δίνονται κονδύλια αν δεν τηρείται η, η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αυτό το λέω εξ αρχή. Μερικέ φορέ μάλιστα μπλοκάραμε σημαντικά έργα για πολλά χρόνια όταν υπήρχαν αμφιβολίε προ την κατεύθυνση αυτή. Να τονίσω επίση ότι τα χρήματα, τα κονδύλια των διευρωπαϊκών δικτύων είναι από τα κονδύλια που παρακολουθούνται όλο εξαιρετικά στενά ερχό, ερχό, ερχόμαστε και σε εσά σε οποιαδήποτε επιλογή κάνουμε από το 2008 και μετά. Και αυτό ήταν μια απάντηση και στην κυρία Μπιλμπάο. Υπάρχει πλήρη διαφάνεια και για τα κριτήρια επιλογή. Δεν υπήρχαν αντιρρήσει εδώ. Έγινε μια ερώτηση για τη μοντελοποίηση. Και εδώ συμφωνώ με τα συμπεράσματα της μελέτης για τα εργαλεία αυτά. Δουλεύαμε χρόνια προσπαθώντας να επενδύσουμε εκατομμύρια και λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα των παραγόντων που παίζουν στον τομέα αυτό δεν είναι δυνατό να υπάρξουν λύσεις ικανοποιητικού χαρακτήρα σε τέτοια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο ετοιμάζουμε ένα δεύτερο μοντέλο που συμπληρώνει τα εργαλεία αυτά και βελτιώνει την κατάσταση. Τελευταία παρατηρήση, πρώτη απάντησή μου. Η απάντηση είναι ότι μαζί με σας ετοιμάζουμε ένα νέο πλαίσιο που αναφέρεται στη μελέτη, περιλαμβάνει μια ισχυρή μεθοδολογία, δίνουμε προτεραιότητε σε βασικά εργαλεία και προτείνουμε την υλοποίηση ε, με τους συντονιστές, διότι αυτό θα γίνει με βάση τους διαδρόμους και θα απαντήσει στα ερωτήματα που δεν μπορούν να τεθούν σήμερα. Πρώτα θα κάνουμε ανάλυση λοιπόν των διαδρόμων και των διαδικασιών υλοποίησης και μετά θα δούμε τι χρειάζεται. Δεν χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, χρειαζόμαστε τις υφιστάμενες ε, δομές, μικρά έργα και τα λίγα μεγάλα έργα που είναι κυρίως διευρωπαϊκά και bottleneck θα επιτρέψουν την υλοποίηση του δικτύου. Ευχαριστώ κύριε Κλάμερ. Η πρόταση της Επιτροπής είναι κρίσιμη και ένα σημείο που θέλω να τονίσω, το έχετε ψηφίσει και θετικά, είναι η απόφαση για τον διάδρομο. Εν τέλει, αυτό που θα μείνει από όλα είναι θα τηρήσουμε την προθεσμία του, 20, του 2030 και αν ναι θα έχουμε τα εργαλεία Η απόφαση είναι απόφαση που μπορούμε να δεχθούμε με τους δύο εισηγητές και περιμένουμε τα κείμενα. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Έχετε 7 λεπτά για να απαντήσετε τώρα σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, γιατί πρέπει στο δεκάμιση να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω. Εγώ. Υπήρξε μια ερώτηση για τους Ευρωπαίους συντονιστές. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και είδαμε ότι η ανταπόκριση ήταν διαφορετική. Εντάξει, κάποιοι είπαν ότι δεν έχουν τις κατάλληλες προφορίες, άλλοι υποστήριξαν πολύ θερμά τα σχέδια, άλλοι μας είπαν ότι υπήρχαν διασυνοριακά προβλήματα και με βοηθούσαν να έχουμε εναρμόνιση των νομοθεσιών. Είναι σαφές ότι είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη τέτοιου είδους σχεδίων και για την πρόθεσή τους. Ε, για την Α11 και επρόκειτο για ένα σχέδιο ε, ανάπλασης, ανακαίνησης του αυτοκινητοδρόμου ε, σε διαφορετικά στάδια, καλύπτοντας ε, διάφορες χιλιομετρικές αποστάσεις ανάλογα με τη χρηματοδότηση του Γερμανικού Υπουργείου Μεταφορών. Καταρχάς χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο, είχαμε προβλέψει 2010 ολοκλήρωση, όμως ολοκληρωθούν ε, τα έργα να το 2014. Στην ε, Σεβίλη, Ουέλβα είχαμε περισσότερες δυσκολίες, διότι δόθηκε μια άλλη προτεραιότητα στη χρηματοδοτή. Και ενδεχομένω να μην έχουν υλοποιηθεί πλήρω γιατί τα άργα δεν ε, σημείωσαν πρόοδο και μέχρι το 2012 υπήρχε συζήτηση να μην ε, οικοδομηθεί το τούνελ, να οικοδομηθεί μια γέφυρα. Τελικά αποφασίστηκε να ακολουθεί ο του τούνελ. Και δόθηκαν και σχετικές συμβάσει στις εταιρείες αλλά οι αρχικές πληροφορίες ε, που λάβαμε ήταν ότι ήταν ε, ολοκληρωμένο το έργο. Μεγάλες διαφορές λοιπόν, εν μέρη και λόγω της οικονομικής κρίσης φυσικά. Για τα καλά έργα νομίζουμε ότι η δεύτερη φάση του West Coast Mainland ήταν ένα καλό τέτοιο έργο. 50 χιλιόμετρα περίπου σε μάκρος. Με διαφάνεια υλοποιήθηκε και σε διαφορά τα Υπουργεία, τους ελεγκτές, τις σχετικές αρχές που εμπλέκονταν. Κάθε χρόνο υπήρχαν σχετικές μελέτες για την πρόοδο του έργου. Και παρά το γεγονός ότι ήταν μεγάλο έργο δεν ξεπεράστηκε το προβλεπόμενο κόστος. Λόγω της καλής συνεργασίας των διαφόρων φορέων. Ένα άλλο στοιχείο, τα κριτήρια για την επιλογή των έργων. Δεν ε, αναζητήσαμε ειδικά έργα με πρόβλημα. Θέλαμε να υπάρχει μια ισορροπία περιφερειακή και φυσικά λόγω του κριτηρίου του μεγέθους είχαμε επιλέξει τέσσερα από τα μεγάλα αυτά έργα τα οποία ήταν σε εξέλιξη και επίσης χρειαζόμασταν και κάποια εξπόστα έργα και γι' αυτό δεν συμπεριλάβαμε το Λιόν, το Ρήνο. Έπρεπε να κάνουμε επιλογές. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Μάλιστα. Για να προσθέσω κι εγώ τις δικές μου απόψεις. Καταρχάς, ε, ακούσαμε την ερώτηση κατά πόσον είναι απαραίτητο να εναρμονιστεί οι διαδικασίες αξιολόγησης. Εγώ θεωρώ ότι ναι, είναι απαραίτητο. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί παντού η διαδικασία, αλλά χρειάζεται μία εναρμόνιση. Ένα παράδειγμα, ή μέθοδοι στη Γερμανία και στη Γαλλία περνάνε αποφάση αναθεώρησης και εκ νέου διαμόρφωσης, αλλά δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση. Και θα έπρεπε και η Επιτροπή να συμμετάσχει, όχι προδιαγράφοντας ε, υποχρεώσεις ε, κατά την αξιολόγηση, αλλά για να συστήσει σημεία αξιολόγησης που είναι σημαντικά για την ποσοτικοποίηση της ε, ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και για την ευρωπαϊκή συγκρισιμότητα. Αυτό για να απαντήσω μία από τις ερωτήσεις σας. Να πω επίσης ότι σέβομαι ιδιαίτερα το έργο των εισηγητών που είναι εξαιρετικό και δεν μας βρίσκει σε τίποτα αντίθετος. Κατά δεύτερον, ποιος είναι ο ρόλος των Ευρωπαίων συντονιστών και των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Το εξετάσαμε το ρόλο των συντονιστών και είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σώμα που θα συντονίζει τις δευτεριότητες και στις δύο πλευρές του διαδρόμου. Και γι' αυτό εκτιμούμε το ρόλο των συντονιστών και θέλουμε να ενισχυθεί, να ενισχυθεί ο ρόλος του. Συμμετοχή των περιφερειών, σημαντικός σε ό,τι αφορά τους εμπλεκόμενους φορείς που θα πρέπει να συμμετάσχουν εξ αρχής. Σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει δυνατότητα να μην συμμετάσχουν οι τοπικοί φορείς είναι πραγματικά δύνατον. Από την αρχή της φάσης του σχεδιασμού. Τώρα πρόβλεψη του αντίκτυπου της κρίσης. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον για τα επόμενα 20, 30, 50 χρόνια. Αυτό είναι σαφές. Αλλά ενώ αυτό ισχύει και για μικρές και για μεγάλες χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να εναρμονίσουμε κάποιες προσεγγίσεις μέσω ενός ενοποιημένου μοντέλου για ένα μελλοντικό σενάριο. Και το έχει πράξει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα χαθεί, για παράδειγμα, λόγω της κρίσης μια ολόκληρη δεκαετία. Και με βάση αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ένα μοντέλο για τη μελλοντική ανάπτυξη των περιφερειών και των χωρών. Ο δοντολογικός κίνδυνος. Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Και γι' αυτό λοιπόν το ποσοστό χρηματοδότησης επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το έργο. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εξ αρχής και θα πρέπει να αποφευχθεί. Ιδάλλως ο σχεδιασμός του έργου δεν θα είναι σωστός και η ανάθεση του έργου θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά. Δεν θα εισέλθω στο θέμα των PPP γιατί είναι διαφορετική η άποψή μου και θα μου πάρει χρόνο να το εξηγήσω. Να σας πω επίσης ότι η σύνδεση μεταξύ της αρισιμότητας και της αναλογικότητας είναι απαραίτητη, γιατί είναι σημαντικό αν η συγχρηματοδότηση είναι 10% ή 60%. Στο 60% η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να ληφθεί πολύ παραπάνω υπόψη σε σχέση με ένα ποσοστό χαμηλό συγχρηματοδότησης. Τελευταίο σημείο, το εργαλείο Trans Tools στο μεγαλύτερο τμήμα της αξιολόγησης χρησιμοποιούμε αριθμητικά στοιχεία του TransTool που δημιουργούνται με το μοντέλο TransTool. Δεν είναι μόνο επιστημονικό λοιπόν το εργαλείο αυτό. Δεν είναι ένα παιχνίδι επιστημονικό, όχι. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την ποσοτική, ε, τον ποσοτικό καθορισμό της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν και πιο απλά εργαλεία. Είναι δύσκολο και περίπλοκο εργαλείο. Μία εβδομάδα παίρνει ένας υπολογισμός και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνουν υπολογιστικές, ε, υπολογιστική εκτίμηση διαφόρων σενάριων και γι' αυτό λοιπόν στην, ε, στην επόμενη φάση θα πρέπει να αναπτυχθούν για να καταστούν πιο αξιόπιστα τα εργαλεία του Trans Tools και να καταστούν και πιο εύκολα στη χρήση τους, προκειμένου να μπορούμε να αναλύουμε πιο, πολλές, πιο πολλά σενάρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο συμμετέχοντες για τις παρεμβάσεις και διότι απάντησαν στις ερωτήσεις τους και η έκθεση που παρουσίασαν όντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τα μέλη. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και συνάδελφοι, θα τα ξαναπούμε το απόγευμα στις 3. Ευχαριστώ.